Allora. Dear colleagues, we can uh, start with a high... Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε με το σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε, αν δεν έχετε ενστάσει, να την εγκρίνουμε, χωρίς τροποποιήσεις. Σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Από την αποστολή μας στο Ελσίνκι έχουμε την αναφορά και τα έγγραφα. Ήταν στις 17 ε, έως 19 Μαΐου. 20 γλώσσες για τη διερμηνία. Και φυσικά είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά τα έγγραφα. Item ε, σημείο 3. Συστάσεις ε, των συντονιστών έχουν κυκλοφορήσει με email. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται αν δεν έχετε κάποιες αντιρρήσεις. Συγγνώμη, πρέπει να επιστρέψω στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Στις 3 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε Τελετή για την υπογραφή της περιβαλλοντικής πολιτικής του 2016 στα πλαίσια του ΕΜΑΣ για την περιβαλλοντική τυποποίηση θα υπογραφεί το έγγραφο από τον πρόεδρο ε, Σούλτσο και από τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου Κλάους Βέλα. Ξέρετε ότι είναι σε θελούσια βάση και ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις ε, βάσει με τον κανονισμό μας και στους τρεις χώρους εργασίας από το Δεκέμβριο του 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία το ΕΜΑΣ και είναι ακρογωνίως ε, λίθος αυτή η πολιτική για την ε, προηγούμενη και την τρέχουσα θητεία. Ε, ε, για το 2016 έχουμε εγκρίνει από τις 9 Μαΐου την αναθεωρημένη μας περιβαλλοντική πολιτική. Παρακαλώ να παρευρεθείτε όλοι στην τελετή υπογραφής της νέας ε, πολιτικής ΕΜΑΣ. Τώρα... 26 Απριλίου, τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης στο σημείο 4 δηλαδή, εγκρίνω τα πρακτικά, δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Αναπομπή για, την, ε, για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις τώρα, σημείο 5. Ε, τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων για, την, για τους επίσημους ελέγχους. Ε, στις 15 ε, Ιουνίου έγινε ο τελευταίος τριμερής διάλογος, σύνολο 17 συσκέψεις σκιωδών και 15 τεχνικές συσκέψεις, 8 μήνες διαπραγματεύσεις με δύο διαδοχικές προεδρίες. Ε, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας. Ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και αύριο θα εγκριθεί επίσημα από την Κορεπέρ και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ θα ψηφιστεί ε, στη συνεδρίασή μας του Ιουλίου. Κυρία Κάντεμπαχ, ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Είναι πολύ καλή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Περνάμε στο σημείο 6 ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπου τη Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή τη νομοθεσία για τα απόβλητα, οδηγία πλαίσια για τα απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασία εφαρμογή περιβαλλοντική νομοθεσία. Θα θυμάστε πως ε, Είχαμε προβλέψει μια πρώτη συζήτηση, η οποία και έλαβε χώρα, όμως δεν μπορέσαμε τελικά να καταλήξουμε θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, δηλαδή ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε απαντήσεις. Ο συνήθως προτείνω να ακούσουμε πρώτα απ' όλα την Επιτροπή και ευχαριστούμε τον κύριο Σαουντάσκας για την παρουσία του. Μετά τις απαντήσεις της Επιτροπής προς τις ερωτήσεις που έχουν προϋποβληθεί θα αρχίσει η συζήτηση με τους συναδέλφους, ε, τα μέλη της Επιτροπής που παρίστανται. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αρχίζουμε με την ε, πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η πρώτη ερώτηση σχετίζεται με τα υποπροϊόντα και τα τελικά απόβλητα, end of waste, σας ευχαριστώ που διοργανώσατε τη σημερινή συζήτηση γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο το ζήτημα και πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Λοιπόν, οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη-μέλη να ερμηνεύσουν σωστά την έννοια των αποβλήτων, να διακρίνουν τι είναι απόβλητο και τι μη απόβλητο στην παραγωγική διαδικασία και στη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Βασιζόμαστε και στην ομολογία. Ε, στα άρθρα 5 και 6 έχουμε τρεις διαφορετικές οδούς ε, σε σχέση με το πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο και εξαρτάται ποια βάση χρησιμοποιείται. Πρώτον, βασόμαστε σε ευρωπαϊκά κριτήρια. Δεύτερον, σε εθνικά κριτήρια και τρίτη εναλλακτική είναι να έχουμε κατά περίπτωση αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά κριτήρια πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει μια άλλη οδηγία, ούτω ώστε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν ότι η εύρυθμη λειτουργία τη ενιαίας αγορά δεν υπονομεύεται από την εφαρμογή τέτοιων εθνικών κριτηρίων. Τα κράτη-μέλη για να θεσπίσουν αυτά τα εθνικά κριτήρια βασίζονται ω επιδοπλίστων στο ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια σε αυτό το τομέα και ε, στο ότι ότι ζητάει η βιομηχανία συγκεκριμένα κριτήρια για ένα κλάδο. Μετά την εφαρμογή τη οδηγία πλαίσιο, τα κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει τουλάχιστον 21 αποφάσει σε σχέση με εθνικά κριτήρια και ε, τα περισσότερα, τις περισσότερες κοινοποίησεις ε, έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο 13, 2 ε, από την Γαλλία, την Αστρία και την Ολλανδία και ούτω καθεξής ε, και σχετίζονται με διάφορα προϊόντα για ανακύκλωση, στερεά απόβλητα, να χρησιμοποιήσει και το καθεξής. Έχουμε εκδώσει λεπτομερείς ε, εκθέσεις ε, για τη διαπίστωση της τυποποίησης εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και μόνο σε μία περίπτωση και πιο συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα κριτήρια σε σχέση με τα επεξεργασμένα έλαια, το, ε, κινήσαμε τη διαδικασία επί παραβάση το πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Ε, εκεί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρίνηση των άρθρων 5 και 6 μέσα από πρόσδοση ενεργού ρόλου και ευθυνών στα κράτη-μέλη για να λαμβάνει αποφάσεις σε δυνάμει αυτών των άρθρων για την ε, βιομηχανική συμβίωση. Δεν προτείνουμε τροποποίηση αυτών των τριών διαφορετικών αλλακτικών λύσεων, δηλαδή ευρωπαϊκά εθνικά κριτήρια και κατά περίπτωση εθνικά κριτήρια, ούτε και προτείνουμε να τροποποιηθούν οι φυστάμενοι όροι, διότι ε, ε, προκύπτουν από την ονομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε λάβει γνώση ε, σημαντικών προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο που θα αιτιολογούσαν μια τροποποίηση των όρων καμιά φορά. Έρχονται σε επαφή με μας επιχειρήσεις σε σχέση με τα υποπροϊόντα και τα, ε, και τα τελικά απόβλητα και για, έχουμε εκδώσει καταθετήριες γραμμές ε, βάσει της νομολογίας και βάσει των πληροφοριών που έχουμε από τα κράτη-μέλη. Ε, και είμαστε πάντως στη διάθεσή τους για περαιτέρω διευκρινήσεις. Για τις μελλοντικές εξελίξεις, για τα κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα θέλαμε να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα που έχουμε παρόλα αυτά. Προτού ε, ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει προσθέμενη αξία για να εκπονήσουμε νέα ευρωπαϊκά κριτήρια. Ε, με προσοχή θα πρέπει να προχωρήσουμε διότι ε, ε, χρειάζονται πάρα πολλοί πόροι για να εκπονεθούν νέα κριτήρια και δεν είχαν τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι στιγμή. Ε, μέσα στο πακέτο τη κυκλική οικονομία προβλέπονται παρόλα αυτά νέα κριτήρια για τα απόβλητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και έχουμε και την αναθεωρημένη πρόταση για τα λοιπάσματα. Οπότε προβλέπονται επιπρόσθετα κριτήρια για τα απόβλητα της καύσης και πυρόλησης. Ε, και ε, στη συνέχεια για τα στερεά απόβλητα έχουμε την περίπτωση της Ιταλίας ε, που κοινοποιήθηκαν τα εθνικά κριτηρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε λεπτομερή σχόλια και λήφθησαν υπόψη για τα εθνικά κριτηρία από την Ιταλία και έτσι μειώθηκε η χρήση των στερεών ανακτημένων αποβλήτων μόνο ε, στα εργοστάσια ε, τα οποία λειτουργούν βάσει της αντίστοιχης οδηγίας και ε, γι' αυτό και εφαρμόστηκαν οι αξίες, οι τιμές που επιτρέπονται από τη συγκεκριμένη αυτή οδηγία για τη διαχείριση των εργοστασίων. Λαβία. Ευχαριστούμε. Απαντήσατε στην πρώτη ερώτηση. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν κάποια προσθήκη. Τόμπας. Uh, ευχαριστώ να ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσει. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το θέμα της, ε, του πόσο συνεκτική είναι η πολιτική της Ένωσης θα συζητήσουμε αργότερα αλλά ακούγοντα την Κομισιόν δεν έχω πιστεί ότι τα κριτήρια τα οποία αναφέρατε για τα τελικά απόβλητα θα οδηγήσουν σε κάποια συνοχή στην πολιτική αυτή. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους από την κάθε χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν δυσκολεύεται να παρακολουθήσει βέβαια το κάθε κράτος μέλος για να βρει λύσεις. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, ε, διαφορετικές προσεγγίσεις. Καλό θα ήταν να εξετάσετε λίγο αυτά τα κριτήρια από χαρακτηρισμού και να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα τελικά. Γιατί τα προβλήματα που έχετε εσείς θα τα αντιμετωπίσουμε και εμείς. μπορούμε να το δούμε αυτό και διμερός, αλλά εάν μπορείτε να διευκρινίσετε, να αποσαφηνίσετε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τα κριτήρια αυτά, θα ήταν χρήσιμο. Πρόεδρος, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω για την ερώτηση. Έχουμε διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια χαρακτηρισμού. Στο χαρτί μπορεί να δίνεται εντύπωση ότι είναι καλά αυτά τα κριτήρια, βοηθούν ε, για την, την ενιαία αγορά, βοηθούν τις επιχειρήσεις, ε, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για μια σειρά από λόγους. Υπάρχουν μια σειρά δηλαδή από γεγονότα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη έχουμε ένα τέτοιο κριτήριο αποχαρτηρισμού για, το, για τα μέταλλα και το γυαλί. Αλλά δεν λειτουργεί. Ε, στην Ιταλία υπήρχε ευτυχώ ένα πανεφερές εθνικό κριτήριο και έτσι λειτουργεί. Αλλού δεν λειτουργεί. Δεν χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για το γυαλί. Θα θυμάστε πριν από μερικά χρόνια είχαμε ένα κριτήριο και για το χαρτί ήταν μια απόπειρα η οποία ε, δεν ευωδόθηκε. Διότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων ε, μεταξύ των ανακυκλωτών και των συλλεκτών. Και αυτό συμβαίνει με τα κριτήρια χαρακτηρισμού. Διότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, κάποια πρότυπα και αυτά τα πρότυπα μπορεί να ικανοποιούν κάποιους αλλά ενδεχομένως ε, να παρεμποδίζει το έργο άλλων. Ή αυτό που μπορεί να συμβεί ή αυτό που συνέβη, με το χαρτί, είναι ότι όταν υπάρχει υπερβολική συλλογή χαρτιού, ε, τότε προκύπτουν προβλήματα και πρόκειται για εντατικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν έχει πραγματικά νόημα να επενδύουμε όταν αυτά τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να εφαρμοστούν στα στις εθνικές αγορές που έχουν τις δικές τους ανάγκες. Έως τώρα δεν έχουμε ακούσει για προβλήματα από τις επιχειρήσεις που να μας πούν δηλαδή ότι χρειάζονται οπωσδήποτε αυτά τα κριτήρια. Κάποιες ενώσεις λένε ότι χρειάζονται κριτήρια, αλλά όταν ρωτάμε τι ακριβώς θέλετε, αυτοί αναφέρουν σε πολύ συγκεκριμένε ανάγκες που έχουν, οι οποίες δεν συνάδουν με τις ανάγκες άλλων. Δηλαδή, αναποκρινόμενοι σε κάποιους, ε, προκαλούμε ζημιά σε άλλου. Προτιμούμε λοιπόν να ελέγξουμε τι κάνουν τα κρατημέλη σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε βέβαια να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γι' αυτό άλλωστε στην τροπημένη οδηγία έχουμε ζητήσει να, να αναφέρεται η δυνατότητα και η υποχρέωση των κρατών μελών ε, για το κριτήριο αυτό, για τα κριτήρια αυτά και να αποφασίσετε ένα περίπτωση έτσι ώστε να μην το κάνουν οι επιχείρησει από μόνε τους. Από εκεί πέρα λοιπόν εμείς ελέγχουμε αν όλα αυτά λειτουργούν καλά, αν συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αν δεν, δεν δημιουργούνται εμπόδια στην αγορά. Τώρα, εάν δούμε το σύνολο του κύκλου των αποβλήτων, ε, η άλλη οδός και αυτό το λένε πολλοί ανακυκλωτές και το κάνουν, είναι ότι παράγουν προϊόντα από τα απόβλητα αυτά. Και στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζονται κριτήρια από χαρακτηρισμού Αυτό που χρειάζεται είναι να συμμορφωνόμαστε άμεσα με, την, με τις απαιτήσει για την πολιτική προϊόντων. Ε, περί υγείας, περιβάλλοντος κτλ. Ε, είναι λοιπόν η πραγματικότητα πιο περίπλοκη και απαιτεί άλλες λύσεις. Εμείς λέμε να μην κλείσουμε την πόρτα στα κριτήρια αποχρητηρισμού. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν. Σας είπα παραδείγματος χάρη ότι είχαμε κάτι σχετικό ε, για τα λοιπάσματα, αλλά κατά τα λοιπά πρέπει να είμαστε αναλογικοί στην προσέγγιση μας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχει άλλο κανείς που να θέλει το λόγο, να περάσουμε στο επόμενο σημείο ευθύνη του παραγωγού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Ίσως είναι μια από τις λίγες επιτυχείς ε, εκβάσεις ε, της πολιτικής μας. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν αυτή η αρχή της εκτεταμένης ε, ευθύνης παραγωγή, του παραγωγού να ισχύσει και στο μέλλον. Είναι σημαντικό αυτό και για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα για την εφαρμοστικότητα της ε, ε, εκτεταμένης ε, ευθύνης παραγωγού στην, στο εμπόριο εξ στην οδηγία πλαίσιο λέμε ότι μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη μορφή ευθύνη στα κρατημέλη προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παράγει, επεξεργάζεται πολύ ή εισάγει προϊόντα. Με τη βάση αυτής της διάταξης τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν την εκτεταμένη ε, ευθύνη παραγωγού ε, προς φυσικά νομικά πρόσωπα που ε, πολλούν, εισάγουν προϊόντα και ανεξάρτητα από το πώς πολλούνται τα προϊόντα οι εθνικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα ε, για να προβούν συγκεκριμένους ελέγχους. Σε ό,τι αφορά τώρα το ηλεκτρικό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσει για τους παραγωγούς ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το εμπόριο εξ αποστάσεως. Η Κομισιόν προτείνει ελάχιστες απαιτήσει. Αυτό τάση οι προδιαγραφές θέλουν να βελτιώσουν τη διαφάνεια των συστημάτων και την παρακολούθησή του, την εφαρμογή από τι αρμόδιε αρχέ και από τι οργανώσει παραγωγών τις ίδιες. Πιστεύουμε ότι αυτό θα δώσει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά το διεθνέ εμπόριο εξαποστάσεω και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των free riders. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα της, του Ιταλικού συστήματος, Υπάρχει ένα μου που λέγεται κονάι το οποίο ε, οργανώνει αυτό το σύστημα. Ε, ε συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, και με την αφορά συσκευασία, ε, διότι οι οδηγίες δεν προβλέπουν συγκεκριμένους κανόνες για, τη, για την χρηματοδότηση. Στην νομοθετική πρόταση τώρα όμως μιλάμε για κάποιες γενικές απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά EPR και, αυτό, και αυτές οι προδιαγραφές θα ισχύσουν και για το Ιταλικό σύστημα Κονάι. Ε, ε, αυτό θα καλύψει όλο το κόστος ε, διαχείρισης αποβλήτων των προϊόντων. Και αυτό θα οδηγήσει, όπως λέει και ο, και ο, και ο Ευρωβουλευτής, σε μείωση του κόστους. Σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες που προτείνονται στο άρθρο 8 του σχεδίου οδηγίας θα έχει τρία χρόνια για την, θέση, για την ε, συμμόρφωση με τις νέους κανόνες μετά την θέση σε εφαρμογή της οδηγίας. Ό,τι αφορά την ε, ε διαδικασία παραβάση που έχει ξεκινήσει, εμείς παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, παρακολουθούμε ότι η Ιταλία σέβεται, ε, και Ιταλία σέβεται τις δεσμεύσεις, έχει ε, δεσμευθεί να εξετάσει τα υπόλοιπα περιφερειακά της σχέδια εντός του 2016 η Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από συναδέλφους για το θέμα αυτό. Όχι. Ωραία. Να περάσουμε στο, στο ερώτημα για τα, ε, τα, επιμέρους quest streams και τις σχετικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ για το θέμα της ε, παράνομης εξαγωγής ε, των ε, οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος κύκλου ζωής. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ. Έχουμε πρόβλημα οικονομικό, διότι έτσι χάνονται πολύτιμοι πόροι. Και ο κύριος Φλόρενς βεβαίω έχει άποψη σημαντική από αυτού. Εμείς επιβεβαιώνουμε την, ε, τις πρώτες εκτιμήσεις ότι περίπου 2,5 με 3,5 εκατομμύρια ε, οχήματα ε, χάνονται, δεν καταγράφονται ούτε ως οχήματα που βρίσκονται στο τέλος ή κύκλου ζωής τους. Μέρος των οχημάτων αυτών δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Πρέπει να θεωρηθούμε ότι παρανόμως λοιπόν έχουν αποσυρθεί τα, αυτο, τα οχήματα αυτά που λείπουν ε, οδηγούν σε έλλειψη πόρων. Ε, παρακάμπτονται οι κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας ε, και βεβαίως και οι κανόνες ασφάλειας εφόσον πολλούνται ως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι κάνουμε από αυτού για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό χρειάζεται δράση σε διάφορα επίπεδα, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιβαλλοντικών και αρχών καταγραφής ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα συστήματα καταγραφής ε, και του εμπορίου των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει πάρει μια πρωτοβουλία από αυτού. θα ξεκινήσει το καλοκαίρι η διαδικασία για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων, να μειωθεί το παράνομο dumping ή η παράνομη ε, μεταφορά οχημάτων στην, ε, στο τέλος κύκλου ζωής. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης αναμένεται στα μέσα του ερχόμενου έτους, ό,τι αφορά τώρα, μάλλον από την 1η Μαρίου του 2016, από φέτος δηλαδή, οι νέε τροπολογίε ε, σε ό,τι αφορά την αποστολή αποβλήτων, ε, ενισχύει τους ελέγχους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προετοιμάζει και εφαρμόζει πράξεις που δημιουργεί έναν πίνακα συσχετισμού έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα τα αγαθά εκείνα τα οποία αποστέλλονται ως απόβλητα ή τα απόβλητα μάλλον που αποστέλλονται ως αγαθά. Ε, Επίση, η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει μια σειρά από καθένα γραμμέ και να βοηθήσει στα κρατημέλια ώστε να μειωθεί η ε, παράνομη ε, αποστολή ε, οχημάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα την, την καύση στην Ιταλία, πρόσφατα είχαμε δύο γραπτές περιβαλλοντικές ερωτήσεις από γερουσιαστές και αυτό Μα ανησύχησε. Θα έρθουμε λοιπόν σε επαφή με τι Ιταλικές αρχέ για να ερευνηθεί το θέμα περαιτέρω. Σε μια πρώτη αντίδραση μπορώ να σα πω ότι κάποιε νέε δυνατότητε καύση μπορεί να χρειαστούν στην Νότια Ιταλία. Το θέμα είναι πόσε Υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα εδώ που τίθενται. Αυτή τη στιγμή ε, φαίνεται ένα κατάλληλο αριθμό ε, της καύσης, κατάλληλα τα ποσοστά 21% το 2014 είναι ένα καλό ποσοστό αν δούμε δηλαδή το σύνολο της χώρας. Και βεβαίω αν αυξηθεί αυτή η προσπάθεια υπάρχει ένα κίνδυνο να δικαιωθούν οι στόχοι που έχουν το 2020, 2025 και το 2030. Επίσης, αυτές οι νέες δυνατότητε αφορούν κυρίως τον νότο της Ιταλίας, όπου είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ε, επένδυση στην ανακύκλωση, σε άλλες μορφές, όπως περιπτώσει, επεξεργασία των αποβλήτων. Θα θέλαμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση ε, το lock-in, ε, δηλαδή το να, ε, αυτά τα απόβλητα να επαγγιδευτούν σε μη κατάλληλες εγκαταστάσεις, διότι αυτό διακυβεύει την όλη προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Now we have a question from Mr. Florence. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από πολλά χρόνια έγραψα την οδικία ως εισηγητής και ήδη τότε μαλώσαμε αρκετά με την Επιτροπή για το ερώτημα ποιος έχει τον τελευταίο λόγο για το αυτοκίνητο. Είναι μόνο ένα χρηστικό αντικείμενο ή είναι ένα σκουπίδι και όλοι αυτοί οι νομικοί στην Κομισιόν δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Μετά υπήρξε διαφωνία με το Συμβούλιο με αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία αυτή δεν λειτουργήσε. Ζω σε, δίπλα σε έναν πολύ μεγάλο αυτοκινητόδρομο από την Αμβέρσα που φτάνει ως πίσω από τη Βαρσοβία από τον οποίο περνούν πάρα πολλά αυτοκίνητα κάθε μέρα τα οποία απορρίπτονται παράνομα στα ανατολικά της Υπήρου μου και όταν σκέπτομαι τι κάναμε στις επιχειρήσεις είπαμε στις επιχειρήσεις πως πρέπει να δημιουργήσουν χώρους απόσυρσης έπρεπε να είναι τόσο οι συνθήκε πρέπει έπρεπε να ήταν τόσο καθαρέ όπω τα σφαγεία. Και στη χώρα μου εκατοντάδε επιχειρήσει έχουν πολύ καθαρού χώρου απόσυρση με πλακάκια εν μέρη έτσι ώστε το λάδι και τα άλλα υγρά να μπορέσουν να αναοροφηθούν με κατάλληλο τρόπο. Και τώρα όλα τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στην Ανατολή ή με πλοία κάπου σε κάποια άλλη ήπειρο. Και με εκπλήσει, με πόση άνεση τώρα εσείς από την Επιτροπή, όχι εσείς προσωπικά αλλά η Επιτροπή, αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα αυτό. Στη χώρα μου χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν απογοητευτεί σπόδρα επειδή οι κανόνες δεν είναι ταιριαστοί. Και όταν ακούω σήμερα πως η Κομισιόν το καλοκαίρι ήδη θέλει να διοργανώσει μια συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων μερών, θα έλεγα ότι αργήσατε πέντε χρόνια. Δεν το εννοώ προσωπικά. Σας άκουσα σήμερα το πρωί με την ησυχία μου. Όλο αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας. Όλη η πολιτική περί αποβλήτων στην Ευρώπη δεν λειτουργεί καλά. Και θα αρχίσω από το πρώτο παράδειγμα. Εάν δεν θα καταφέραμε καν να έχουμε έναν όρο, έναν ορισμό για το τι είναι η ανακύκλωση, όταν έχουμε 5 6 ή 7 διαφορετικές τοποθετήσεις στην Ευρώπη σχετικά με αυτό, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει τότε. Στη θέση της Κομισιόν δηλαδή θα ασχολιόμουν σοβαρά με το ζήτημα και θα σκεπτόμουν τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Ποιος αποφασίζει εκεί έξω για τα παλιά αυτοκίνητα, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο, ποιος ευθύνεται. Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, δεν υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης και οι παράνομοι στην Ευρώπη γελούν για μας. Πάτε μια φορά στην ακτή Εκεί θα δείτε πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα μεταφέρονται εκεί παράνομα. Είμαι αγανακτισμένος, επειδή μιλούμε για μια τεράστια οικονομική απώλεια. Τώρα σε λίγο τελειώνω. Και εμείς με την συνάδελφο Μποναφέ, η οποία προσκόμισε μια πολύ καλή έκθεση, κάνουμε, προσποιούμαστε, σαν να μας ενδιαφέρει η κυκλική οικονομία. Και έχουμε μια τόσο μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό, από όπου διαραίουν οι πρώτες ύλες, και τι κάνει η Κομισιόν, σχεδιάζει το καλοκαίρι μια συνεδρίαση ενδιαφερόμενων μερών. Συγγνώμη, συμμετείχα τότε όταν γράφτηκε το εγγραφό αυτό. Δεν ήσασταν τότε ακόμα στην Κομισιόν, μαλώναμε συνέχεια με την Κομισιόν. Έχω τα ονόματα ακόμα. Όχι, ήθελαν ένα πολύ φιλελεύθερο έγγραφο που είχε ως αποτέλεσμα σήμερα από χίλιες τρύπες να μας ξεφεύγουν οι πρώτες ύλες και να εξάγονται. Οι άλλοι γελούν με μας και εμείς είμαστε χαζοί. Ευχαριστώ πολύ. Άλλε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Όχι. Τότε δίνω τον λόγο και πάλι στην Επιτροπή. Το σχολείο σας. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με την κριτική ανάλυση του κυρίου Φλόρεντς Φυσικά πρέπει να προσέχουμε. Αυτό είναι μια οδηγία. Όταν ρωτάτε για το ποιο είναι αρμόδιος για την εκτέλεσή της, γνωρίζουμε είναι τα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν για το κατά πόσον εκτελούν ή όχι την οδηγία αυτή. Αφετέρου, δεν θα έλεγα ότι υπήρξε πλήρης αποτυχία. Αν κοιτάξει κανείς τους βαθμούς ανάκτησης εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, πιστεύω πως είναι από τους υψηλότερους μεταξύ όλων των προϊόντων. Συζητήσαμε και πριν για την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί το σύστημα, επειδή το σύστημα ευθύνης του παραγωγού για τις πωλήσει αυτοκινήτων και για την ανάκτηση φαίνεται να λειτουργεί καλά όταν η επιβολή της νομοθεσίας γίνεται με κατάλληλο τρόπο. Το πρόβλημα είναι με τα αυτοκίνητα που λείπουν, τα οποία δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται. Ναι, είναι ένας τρομακτικός αριθμός, είναι εκατομμύρια. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με αυτά. Μπορεί να μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από συναρμολογούνται, επίσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν αποσυναρμολογούνται σε μη ρυθμισμένες συνθήκες δημιουργείται μια στρέβλωση, του ανταγωνισμού για αυτούς που τηρούν την ομοθεσία. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη και ιδίω με τις αρχές ταξινόμησης και διαγραφής των οχημάτων. Έχουμε δηλαδή μία έλλειψη εφαρμογής. Δεν θα έλεγα πως η εξαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι κάτι κακό γενικώς πιστεύω πως αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο αλλού, ας είναι. Φυσικά το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν όντως φτάσουν το τέλος του κύκλου ζωή, ζωής τους και κατά πόσο να αποσυνεργολογούνται με κατάλληλο τρόπο. Η δυσκολία όμως είναι η, η, παράνομη μεταφορά των οχημάτων αυτών που απλά εξαφανίζονται από τις αγορές μας. Τότε συμφωνώ πρόκειται για μια κακή χρήση πόρων, η οποία είναι πολύτιμη. Καθώς περιλαμβάνονται στα αυτοκίνητα, έχουμε πολλές πολύτιμες αλλά και επικίνδυνες ουσίες στα αυτοκίνητα. Εφόσον αποσυναρμολογούνται στην Ευρώπη σύμφωνα με τους κανόνες, τότε όλα πάνε καλά. Αλλά όταν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την κοινωτική νομοθεσία, τότε έχουμε ένα πρόβλημα διαρροής πόρων. Θέλουμε να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να βρουν το μέγεθος, την κλίμακα του προβλήματος και να δούμε αν κατά πόσο μπορούμε να τα καθοδηγήσουμε και να τα παρακολουθούμε πολύ περισσότερο για να διασφαλίσουμε πως η εκτέλεση της οδηγίας αυτής είναι η κατάλληλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο πάλι στον κύριο Φλόρεντς και μια ερώτηση ακόμα. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί, εάν με πολιθεί στην Ανατολική Ευρώπη, δεν μπορώ να πω παρά ωραία, πολύ ωραία. Εάν το αυτοκίνητο είναι εντάξει, αν λειτουργεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ας υποθέσουμε τώρα, λέτε, αναφέρεστε στην ευθύνη των παραγωγών. Τότε συμμετείχα και λέγαμε πως βρήκαμε τη λύση. Γνωρίζετε ποια είναι η ευθύνη των παραγωγών στα ηλεκτρονικά απορρίμματα και στα απορρίμματα αυτοκινήτων. Είναι πολύ απλό. Είστε ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων που αγοράζει μίζες, μπαταρίες και τα λοιπά στην Bosch. Τότε η Bosch καλύπτει τα έξοδα τη διάθεση των απορριμμάτων. Στο τέλος οι Mercedes και οι Audi δεν, δεν ξοδεύουν ούτε λεπτό. Ακόμα και αυτός που κατασκευάζει μια μικρή βιδούλα, ένα μικρό ελαττήριο, αυτός πρέπει να πληρώσει το μερίδιό του στα έξοδα διάθεση απορριμμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μεγάλε επιχειρήσει να μην πληρώνουν απολύτω τίποτα και δεν φέρουν καμία ευθύνη. Δεν την νιώθουν αυτή την ευθύνη. Υπάρχει εδώ ένα κενό. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Και πιστεύω πω η Κομισιόν θα τα καταφέρει. Υπάρχει ένας κατασκευαστής από κυβότια ταχυτήτων, η ZF, η οποία πληρώνει όλη την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η Audi, η Porsche δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Αυτό δεν είναι ευθύνη παραγωγών. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και όταν δεν υπάρχει ευθύνη παραγωγών, τότε μας ξεφεύγουν τα εμπορεύματα. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση τώρα. στον αυτοκινητοδρυμο α Α40 που περνάει το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, συνεχίζει στην Πολωνία, ποιος ελέγχει, τι μεταφέρουν τα φορτηγά αυτά. Θα ήθελα να το ξέρω. Αν μπορέσετε να ανατρέψετε την απόψή μου θα είμαι ικανοποιημένος, αλλά φοβούμαι ότι δεν γίνεται. Ε, um, τα κράτη-μέλη μπορούν να ερμηνεύσουν ε, διαφορετικά ε, την ευθύνη αν πρόκειται για βιομηχανία που παράγει αυτοκίνητα ή για κάποιον που τα διαθέτει στην αγορά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετική ε, η κατάσταση στη Γερμανία που παράγει από το των αυτοκίνητα Κανένας δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη ε, και τα, οι γερμανικές αρμόδιες αρχές ε, θα πρέπει ε, να εφαρμόσουν την νομοθεσία και να αποδώσουν ευθύνες. Φυσικά υπάρχουν κίνητρα, μια ένας άλλος μεγάλος κατασκευαστής σε κάποια άλλη χώρα έχει έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ε, σύστημα για την επαναπόληση ανταλλακτικών που ε, τα επισκευάζονται και επιστρέφουν στα αυτοκίνητα σαν καινούρια και νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση ένα τέτοιο σύστημα. Ποιος ελέγχει τα φορτηγά τώρα, με ρωτήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, λόγω της ενιαίας αγοράς. Φυσικά αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές. Σε διασυνοριακές περιπτώσεις όμως ε, είναι τα τελωνία υπεύθυνα. Και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τις τελωνιακές αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ε, χάρη στον αναθεωρημένο τελωνιακό κώδικα ε, φυσικά μόνο σε ανταλλακτικά μπορεί κάποιος να το στείλει με, με, με, μεταφορική εταιρεία το αυτοκίνητο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη. Πάντως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε να, είναι να επιστήσουμε την προσοχή των τελωνιακών αρχών, τόσο ώστε μη εγκεκριμένοι μεταπολιτές να μην μπορούν να κάνουν τέτοιες εξαγωγές. Όμως σίγουρα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Λαβία, σας ευχαριστούμε. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 ανώτατα όρια καταλήπων για την ουσία τριακλοπρίντ μέσα υπάνω σε ορισμένα προϊόντα. Η η που έχει εκφράσει τις εντηρήσεις ε, θα ε, πάρει το λόγο. Η κυρία Γκοντίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για τα ανώτατα όρια καταλήγων για την ουσία τριακλοπρίτη στο μέλι. Είναι ένα ζυζανιοκτόνο από τα νέο νοικοτινοειδή. Ένα λεπτάκι γιατί δεν, δεν με ακούω καλά. Τι έλεγα. Είναι ζυζανιοκτώνα από την κατηγορία των νεονικοτινοειδών ε, και ε, διέπεται από την οδηγία για τα μερικά νεονικοτινοειδή. Ε, από το 2013 και 2014 βλέπουμε τριπλασιασμό της κατανάλωσής του, όμως βλέπουμε και αύξηση 31% ολόκληρης κατηγορίας την ίδια περίοδο. Το 2005 δόθηκε η άδεια και η ανανέωση τώρα μελετέται από την ΕΦΣΑ την Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων και Χρησιμοποιείται και για την άθεση και οι μέλισσες εκτίθενται ιδιαίτερα σε αυτή την ουσία μας. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τετραπλασιάσουμε την, ε, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο στο μέλι και γι' αυτό έχω υποβάλει την αντίρρηση. Οι οδηγίες και οι κανονισμοί που καλύπτουν και την χορήγηση της άδεια και τον προσδιορισμό των ενότατων όριων καταλήπων έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τα ζώα και για τους ανθρώπους οι επιπτώσεις ε, για το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και είναι ένας μόνο από του παράγοντες. Επίσης, μας εκπλήσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, παρά όλες αυτές τις ενδείξεις που έχουμε και που μας οδηγούν σε, στην ανάγκη να δείχνουμε σύνεση, διότι υπάρχουν ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, ε, οι οποίοι δεν λειτουργούν βάσει των μελετών σωστά μετά την έκθεση σε αυτή την ουσία. Και έχει επίσης, υπάρχουν υποψίες ότι είναι καρκινογόνος και το μπορεί να αποβεί τοξική σε μεγάλη συγκέντρωση ε, είναι ε, μεγάλος ο κίνδυνος της υγείας ε, λοιπόν με τη χρήση αυτών των ε, ζυζανιοκτώνων, ε, κυρίως στον τομέα της ε, μελισσοκομείας, γιατί πέρα από τα προβλήματα που έχουν ούτως ή άλλως οι μελισσοκόμοι, νομίζω θα εκτεθούν σε αυτόν το περιττό επιπρόσθετο κίνδυνο. Ο κύριος Ανδρουκαίτης, ο αρμόδιος επίτροπος, μας μίλησε εξάλλου για τους κινδυνούς, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και νομίζω μετά τη δήλωσή του θα θεωρήσετε ότι είναι βάση μία αυτή η αντίρρηση που έχω υποβάλει. Η Γερμανία, η συγκήτρια χώρα, έχει εκδώσει μία γνωμοδότηση, η οποία όμως βασίζεται ε, αποκλειστικά και μόνο σε δύο μελέτες. Δεν πιστεύω ότι είναι αμερόληπτη, ε, διότι δεν ε, εξετάζει διαφορετικές καλλιέργειες. Πρώτο πρόβλημα και δεύτερον, το πρωτόκολλο που προβλέπεται κανονικά προβλέπει ε, δύο διαφορετικά ζυζανιοκτώνα, τη χρήση δύο διαφορετικών ζυζανιοκτώνων τουλάχιστον, το οποίο δεν ε, τηρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και πέρα από την ε, τριακλοπρίτε υπάρχουν και άλλες ουσίες και σας παραπέμπω στην γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ για τη, της 23 Φεβρουαρίου για τα ανώτατα όρια καταλήπων ΜΡΕΛ. Ε, τονίζεται εκεί ότι υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει να σου οδηγούν σε γρήγορση... διότι υπάρχουν και οι επιπτώσεις στα ίδια τα ζώα στις μέλισσες η τροποποιημένη γνωμοδότηση ε, του, της ΕΦΣΑ ε, βασίζεται και στον αναθεωρημένο κανονισμό 546 του 2016 για τις εμέλησεις. Θα πρέπει ε, να αναλυθούν λοιπόν τα αποτελέσματα διότι δεν είχαμε στοιχεία στη διάθεσή μας μέχρι τη, τώρα για την μελοσοκομία και προσωμιάζεται με ένα προϊόν πλούσιο σε ζάχαρη το μέλι, κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε και βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν και άλλοι παράγοντε υπόψη, γιατί αλλιώ επηρεάζονται τα αποτελέσματα τη μελέτη. Δεν ε, έχουν διεξαχθεί απαιτούμενε μελέτε, διότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για το τριακλοπρίτ και τι επιπτώσει που έχει στι μελέτε, ακόμη και σε χαμηλή συγκέντρωση. Πλήττεται το νοσοποιητικό των μελισσών ε, κατά τη διάρκεια. Ε, ε, κατά τη διάρκεια της άνθησης και κατά τη διάρκεια της παραγωγής του βασιλικού πολτού ε, και των λιμφών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τετραπλασιασμό του τριακλοπρίτ ε, ο ΕΦΣΑ από το 0,05% προτείνει να περάσουμε στο 0,2% για την περιεκτικότητα τριακλοπρίτ στο μέλι. Δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό με τη βάση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία δεν ισχύει αυτό όμω μέσα στην νέα γνωμοδότηση του ΕΦΣΑ. Εξάλλου αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τον ΕΦΣΑ. Επίση δεν τηρείται η αρχή τη ε, πρόληψη ε, και ε, χρειαζόμαστε αυστηρότατη νομοθεσία. Ο περιορισμό του τριακλοπρίτ στη ΣΥΠΑ είναι μια πραγματικότητα. Είναι μηδενική η ανοχή του τριακλοπρίτ μέσα στο μέλι. Οι ενώσει προστασία των μελισσών έχουν συλλέξει υπογραφή έχουν φτάσει στο μισό εκατομμύριο για να καταλάβετε ποια είναι η άποψη των μελισσοκόμων. Ε, ε τέλος, αυτό το σχέδιο απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας βρίσκει αντίθετο ε, και σας ζητώ να με στηρίξετε γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον μα χωρί μέλισσες. Ευχαριστούμε, κύριο Μπουζόη. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αυτοί οι συνάδελφες, θα ήθελα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα από τους συναδέλφους ΣΥΜΒΕ και τη θέση μας σε σχέση με την πρόταση της κυρίας ε, Γκοντίν. Ο, η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβλέπει ανώτατο όριο καταλήπων για την εργό ουσία τριακλοπρίτε μέσα στο μέλι. Αυτό το MRL ε, θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη για προϊόντα φυτοπροστασίας να χορηγούν άδειες για τέτοιες καλλιέργειες όπου ε, ναι. όπου υπάρχουν μέλισσες είναι ευρύτατο του στο ζυζανιοκτόνο και είναι αποτελεσματικότητα, ε, αποτελεσματικότατο για τα τελευταία 15 χρόνια και βοηθά ε, τις, ε, τους καλλιεργητές ε, διαφόρων ε, καλλιεργειών όπως ποροκυπευτικά ή ελαιούχους σπορούς. Είναι εξαιρετική η λύση του κλειοπρίντε για την διαχείριση των ζυζανίων και για την, πρέπει να διαπιστώσουμε επίσης ότι για την παραγωγικότητα για την εντατική καλλιέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικά τέτοια ζενιοκτώνα, διότι με στοχευμένη χρήση μπορούν να προστατεύσουν την... Ε, τι καλλιέργειέ του από τέτοιου επιβλαβεί ε, οργανισμού. Επίση, ε, ο κανονισμός 1107 του 2015 προβλέπει την θέση σε εμπορία αυτών των προϊόντων ε, όπου βλέπουμε ότι εγκρίνονται προϊόντα που δεν έχουν ε, ε, επιπτώσεις στις μέλησες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Και έτσι έχει κρυθεί ως τέτοιο προϊόν το ζυζανιοκτόνο που περιέχει τριακλοπρίντα από τον ΕΦΣΕ και έτσι διαπιστώνεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των μελισσών όταν γίνεται σωστή χρήση του προϊόντος ε, με συμμόρφωση με τους ε, προβλεπόμενους όρους ε, χρήσης. Πριν από 15 χρόνια έχει να χρησιμοποιείται το 3 κλοπρίν και έκτοτε δεν υπάρχουν αποδείξεις σε σχέση με επιβλαβείς επιπτώσεις για τους ανθρώπους ή για τα ζώα όταν γίνεται σωστή χρήση του προϊόντος. Στη Γερμανία βλέπουμε ότι εντάσσεται στην κατηγορία V2, V2 και άρα δεν είναι χαμηλή η τοξικότητα σε σχέση με άλλα ζενιοκτώνα για τις μέλισσες. Ο ΕΦΣΑ κατέληξε επίσης στο ότι ο προσδιορισμός του ανώτατου όριου καταλήπων MRL για το 0,15 ή 0,2 μιλικρά το ε, κιλό για το τριακλοπρίντε στο μέλι δεν οδηγεί σε έκθεση των καταναλωτών σε ε, τιμές ε, που υπερβαίνουν ε, τις προβλεπόμενες τιμές για την τοξικότητα και άρα δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, λέει ο κ. Σελίμωβιτς, να εκφράσω την εμπιστοσύνη στο σύστημα ασφάλειας και στις επιστημονικές αξιολογήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Θέλω να θυμίσω τα εξής. Στις 18 Φεβρουαρίου η ΕΦΣΑ παρουσίασε την αξιολόγησή της για το τριακλοπρίντ και τα MRL και έφτασε στο συμπέρασμα ότι το προτινόμενο ανώτατο όριο 0,15 ή 0,2 στο μέλη, δεν θα οδηγήσει σε έκθεση σε κίνδυνο ε, του καταναλωτή πέρα από τις τοξικολογικές ε, τιμές αναφοράς, οπότε δεν δημιουργείται κίνδυνος ε, για την υγεία του καταναλωτή. Μετά τη γνώμη της ΕΦΣΑ, η μόνιμη επιτροπή για τα φυτογενομικά 14 ε, με 16 Απριλίου ψήφισε θετικά στο να τεθεί το MRL στο 0,2 με ευρία πλειοψηφία 26, 26 μέλη ψήφισαν, κάτι μέλη ψήφισαν υπέρ. Ε, επίσης στη Γερμανία η ενεργή ουσία δεν θεωρείται επιζήμια ε, για τις μέλισσες. Στη κατηγορία Β4 έχει το υψηλότερο ποσοστό στη Γερμανία και μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές προϊόν. Έτσι λοιπόν το τριακλοπρίντ ακολουθεί μια αργή διαδικασία έγκρισης. Τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Χημική Υπηρεσία, από, την, από τις αρχές ασφαλείας των τροφίμων, τις αρχές των κρατών μελών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι μόνο τα προϊόντα, τα, φυτοπροστατευτικά, τα οποία είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφόσον χρησιμοποιηθούν με βάση τη χρήση που προβλέπεται, ε, μπαίνουν στην αγορά της Ένωσης. Από αυτής της βάσης, είναι ασαφείς ε, οι, λόγοι για αυτό το ψήφισμα και πιστεύουμε ότι πρέπει να απορριφθεί. Ευχαριστώ κύριος Φλόρενς. Um και εγώ ανησυχώ για τις μέλισσες. Αλλά αυτή η ανησυχία κάπως αποσπά την προσοχή από την χρήση νέων νοικοτινοειδών και τους τομείς χρήσης τους. Ας πω ένα παράδειγμα προσωπικό δικό μου. Είμαι καλλιεργητής κράμβης. Τα σποράκια της κράμβης επικαλύπτονται με μια στρώση τόρφης. Εκεί μέσα υπάρχουν νοικοτινοειδή. Ποιο από αυτές τις τέσσερις ομάδες δεν έχει σημασία καταρχήν. Αλλά εκεί υπάρχουν νοικοτινοειδή. Με αποτέλεσμα και εκεί διαφωνώ με τον προλαλήσαντα είναι μια μόνιμη καταπολέμηση εντόμων από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Μαΐου. Πριν από δέκα χρόνια ψεκάζαμε. Τα έντομα πέθαιναν και μετά από τρεις μέρες ξαναέρχονταν. Τώρα έχουμε μια μόνιμη καθημερινή καταπολέμηση εντόμων επί μήνες και θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο δρόκτημά μου Εκεί στους αγρούς της Κράμβης επικρατεί σιγή νεκροταφείου. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε έντομα, ούτε μέλισσες. Έχουν πεθάνει όλα. Δηλαδή αυτό το, αυτή η ουσία είναι διαολεμένη. Δεν ξέρω άμα είναι τοξική, σίγουρα είναι τοξική για όλα τα μικρά ζωάκια που πετούν εκεί δεν έχουμε πλέον έντομα που γίνουν στο υπέδαφος. Έχουμε ζώα τα οποία έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, επειδή έχουν πεθάνει της πείνας, επειδή οι φασιανοί και τα άλλα ζώα δεν έχουν πια να φάνε. Επικρατεί σιγή νεκροταφείου. Και εδώ και κάποια χρόνια σταματήσαμε εθελοντικά εμείς με, το, με την ουσία αυτή και ας με εξηγήσουν οι συνάδελφοι. Εάν χρειάζεστε το, την ουσία αυτή για την κράμβη, το αμφισβητώ. Μπορείτε να περάσετε με ένα συμβατικό μέσο μία φορά τον Αύγουστο και μία τον Σεπτέμβριο, το τα φυτά είναι τόσο δυνατά που δεν χρειάζονται περαιτέρω προστασία. Εκεί την πάθαμε από τη βιομηχανία. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην εκλογική μου περιφέρεια, το όνομά της αρχίζει με B, σκέφτεται πως τέτοιες ουσίες που δρούν επί μήνες πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να κάνουμε τη βιομηχανία να πρέπει να δράσει με θετικό τρόπο, δηλαδή να παρασκευάζει προϊόντα τα οποία δεν θα μολύνουν τα ύδατα. και δεν θα καταστρέφουν τα πάντα επί μήνες. Τα νέα νοικοτινοειδή στο δικό μου αγρό απαγορεύονται εδώ και χρόνια και η σοδιά μου έμεινε όπως ήταν. Για μένα απαγορέψτε όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να πάρει τον λόγο, αλλιώς τον λόγο έχει από την Επιτροπή ο κύριος Φλούεν. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα να εξηγήσω σύντομα πως πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της έγκρισης προϊόντων φυτοπροστασίας και του προσδιορισμού μέγιστων επιπέδων καταλήπων. Όσον αφορά το θηριακλοπίτ, θεωρώ πως είναι σημαντικό να πω μερικά πράγματα. Το θηριακλοπίτ και τα νέα νοικοτινοειδή είναι εγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2005. Η έγκριση λίγη του χρόνου τον Απρίλιο, στις 30 Απριλίου 2017 εγκρίθηκε χωρίς περιορισμούς η μέτρα μετριασμού κινδύνου. Όταν μια τέτοια ουσία εγκριθεί, τότε απόκειται στην ευθύνη των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα προστασίας κατά των δραστικών ουσιών. Μπορούν να ληφθούν μέτρα για τις μέλισσες, παραδείγματο χάρη ε, τα εντομοκτώνα μπορούν να είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες. Μπορούν να χρησιμοποιούνται επί συγκεκριμένε ώρες της ημέρας ή χρονικές περιόδους του χρόνου. Για κάθε έγκριση, τα κράτη-μέλη πρέπει να προσδιορίσουν ένα μέγιστο επίπεδο καταλήπων. Είναι αρμοδιότητα των κρατών, η αξιολόγηση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και της ΕΦΣΑ Επίσης θέλω να τονίσω πως περιορίσαμε δραστικά τη χρήση τριών νέων νοικοτινοειδών το 2013 Είχαμε επιστημονικά στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι τρεις ουσίες αυτές ήταν βλαβερές για τις μέλισσες. Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, το θριακλοπίτ βρισκόταν ήδη στην αγορά αλλά η Κομισιόν με βάση μια δήλωση της ΕΦΣΑ αποφάσισε πως το θιακρολοπίτ και ένα άλλο νέο ήταν χαμηλότερης τοξικότητας, οπότε δεν έπρεπε να συμπεριμπεθεί στον περιορισμό που ίσχυε για τα νέο νοικοτινοειδή. Όπως είπα, η άδεια θα λήξει τον Απρίλιο του 2017. Η διαδικασία ανανέωσης πραγματοποιείται επί του παρόντος από τον εισηγητή, τα κράτη-μέλη και την ΕΦΣΑ. Οπότε τώρα θα ήθελα να φτάσω και στους ενδοκρινικούς διαταρακτές. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση για την οποία εφαρμόζονται μεταβατικά κριτήρια. Όπως είπε και ο Επίτροπος στην περασμένη εβδομάδα απευθυνόμενο στην ΕΦΣΑ και στην ΕΚΑ να προετοιμαστούν για εκθέσεις σχετικά με ουσίες για τις, οι οποίες είναι δυνητικοί ενδοκρινικοί διαταρακτές. Αυτή η εργασία συνεχίζεται και όπως είπα τον Απρίλιο του χρόνου λίγη η άδεια. food. Ο στόχος των ανώτατων ορίων καταλήπων είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων. Τα ανώτατα όρια καταλήπων δεν υπάρχουν για να προστατεύουν τις μέλισσες. Είχαμε πρόσφατα μια δικαστική υπόθεση βάσει μιας νομικής γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν η υπόθεση αυτή αποσύρθηκε από το δικαστήριο. Μας ζητήθηκε να θεσπίσουμε ανώτατα όρια καταλήπων. Για την συγκεκριμένη περίπτωση του Φριακλοπίτ, το ανώτατο όριο καταλήπων μειώθηκε στο, στα 0,05 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Αυτό έγινε λόγω διοικητικής επισκόπησης επειδή τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη δεν υπέβαλαν τα δεδομένα για την ουσία αυτή. Η μείωση του ε, κατώτατου επίπεδου καταλήπων στα 0,5 μιλιγκράμμ δεν οφειλόταν σε ανησυχίες για την ασφάλεια. Εάν διατηρούσαμε το επίπεδο αυτό, τότε τα κράτη-μέλη θα το... δεν θα μπορούσαν να συμφω... συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα επίπεδα και κάποιες ουσίες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πλέον. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη προσέγγισαν την Κομισιόν, κυρίως η Γερμανία, αλλά και άλλα κράτη-μέλη, που έχουν καλή φήμη όσον αφορά τα μελισσοκομικά και ζήτησαν να μειωθεί το ανώτατο αυτό. Η Γερμανία επέβαλε νέα δεδομένα τα οποία αξιολογήθηκαν από την ΕΦΣΑ και δικαιολόγησαν την θέση του ανάδοτου ορίου καταλήπων στα 0,2 μιλιγκράμμ. Αυτή είναι η πρόταση η οποία βρίσκεται επί τραπέζης. Επίσης είχαμε αιτήματα από ενώσεις μελισσοκόμων να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Κατά την αξιολόγηση των ανώτατων ορίων καταλήπων και του αντίστοιχου φακέλου, η ΕΦΣΑ πάντα εξετάζει επίσης την έκθεση στις ουσίες αυτές, ιδίως εκ μέρους ευάλωτων ομάδων. Αυτή λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των ανώτατων ορίων καταλήπων δεν λαμβάνουν υπόψη άμεσες και οι έμεσε συνέπειες για μέλησες. Όπως είπα πριν, αυτό δεν είναι ο σκοπός της νομοθεσίας. Καθώς υπάρχει πλήρης κάλυψη από την νομοθεσία περί ουσιών. Όπως είπα, η πρότασή μας υποστηριχθήκε από πολλά κράτη-μέλη. Είχαμε μόνο δύο αποχές και η Κομισιόν είναι της άποψης πως με το σχέδιο δεν υπερβήκαμε τις εκτελεστικές μας αρμοδιότητες ούτε το πεδίο ισχύω της νομοθεσίας όσον αφορά τη θέσπιση μέγιστων επιπέδων καταλήπων. αλλά και την νομοθεσία σχετικά με την εμπορική κυκλοφορία προϊόντων φυτοπροστασίας. Ευχαριστούμε. Να κλείσουμε εδώ με αυτό το σημείο, να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια, την κυρία Γκοντά. Θα ψηφίσουμε, παραλαμβάνω, σήμερα το απόγευμα στην ΕΝΒΗ και στην Ολομέλεια του Ιουλίου, εφόσον εγκριθεί βεβαίως σήμερα εδώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι οι οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του αποτυπώματος άνθρακα. Είμαστε στην τέταρτη φάση του ETS και επ' αυτού του σημείου έχουμε το σχέδιο κειμένου του εισηγητή και θα δώσω αμέσως το λόγο, θα δώσω αμέσως το λόγο για να μας εξηγήσει τη θέση του και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Ντάνκαν, έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω ε, τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα στον Ηνωμένο Βασίλειο και να πω δύο πράγματα μου επιτρέπετε. Πρώτον, εάν όντως το Ανωμένο Βασίλειο τελικά ψηφίσει ε, ε, το Brexit, τότε θα πρέπει να παραιτηθώ ως εισηγητής. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό το αντιλαμβάνεστε. Δεν θα έχει νόημα ε, και θα συνεχίσει κάποιος συνάδελφος τον οποίο εύχομαι καλή τύχη. επίσης θα πρέπει ο επόμενος συγητής να έχει ένα περιθώριο ευρύ για να μπορέσει να δράσει είναι μια λογική προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, να δώσει την ευκαιρία να ξανανοίξει το φάκελο από την αρχή. Ε, είναι δύσκολο να μας μιλάει κάποιος γερμανικά όταν δεν καταλαβαίνουμε γερμανικά. Εγώ ε, δεν νομίζω ότι θα ψηφίσουμε για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό όμως είναι να το αναφέρουμε αυτό. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Πέμπτης, θα είναι πολύ, ε, πολύ σφιχτό το αποτέλεσμα και τα πράγματα δεν θα είναι όπως το παρελθόν. Και είναι κρίμα που το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης δεν έχει πάρει κάποια μεγαλύτερη έμφαση στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, όλα αυτά πρέπει να είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία, ε, εγώ είμαι απογοητευμένο. Έχω κάνει λόμπινγκ εδώ καιρό για το κοινό ηλεκτρικό δίκτυο. Αν σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό, αυτό θα μπορούσε να παίξει θετικό ρόλο και στη συζήτηση ε, για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό δεν συνέβη. Να μιλήσω τώρα για την, για την έκθεση. Η έκθεση είναι μια απόπειρα να εξασφαλίσουμε ότι θα, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και τις φιλοδοξίες μας. Στο δεν περίμενα εγώ ότι θα φτάσουμε στο 1,5 βαθμό Κελσίου ως αποτέλεσμα. Ε, και αυτό είναι ε, θετικό ότι το πετύχαμε. Αλλά η πρόκληση μπροστά μας τώρα είναι να γνωρίσουμε ότι ευρύτερα ε, δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το προβλήματα με το ETS και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Οι στόχοι του 2030 θα πρέπει να, να Θα πρέπει να δούμε τις φιλοδοξίες μας σε όλες τις προσπάθειες μας Ιδάλλως δημιουργούμε μεγάλε προσδοκίε προσδοκώντα από μια πολιτική να λύσει όλα τα προβλήματα, κάτι που δεν γίνεται στην πράξη και θα ήταν κρίμα να, διαψευθούν οι προσδοκίε ή ήδη Η ίδια η έκθεση περιλαμβάνει καποιε πτυχέ οι οποίε δεν είναι και τόσο δημοφιλεί, Κάποιε άλλε είναι δημοφιλεί, έτσι ε, είναι αυτά. Δεν αμφιβάλλω ότι θα υπάρξουν ε, τροπολογίες, θα υπορθουν τροπολογιε τροπολογίες, 5-6 αναμένω, ε, κάποιο θεωρεί Κάποιοι θεωρούν ότι ε, υποτιμώ ε, τον αριθμό. Ε, εν πάση περιπτώσει όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ να εξετάσουμε το θέμα αυτό λεπτομερώς και να καθορίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, θα έλεγα ότι προσπάθησα να είμαι γαλήνιος, προσπάθησα να είμαι ειλικρινής, ανοιχτός. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση έχει αυτή τη μορφή. Γι' αυτό δεν έχουν γίνει και οι προσαρμογές. Ε, δεν είναι επειδή δεν είμαστε υπέρ ε, ότι δεν είμαστε φιλόδοξοι, μπορεί να, προσαρμοστεί, να προσαρμοστούν οι, οι, οι μας. Τώρα, αν διαφωνείτε, ε, μπορούμε να φανούμε πιο φιλόδοξοι και να τροποποιήσουμε το κείμενο, αλλά δεν νομίζω να βρεθεί απαραίτητη πλειοψηφία για να συμβεί αυτό. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι αναφέρθηκα ε, σε τρία σημεία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να θεσπιστούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καταρχήν, ε, εάν μειώσουμε στο 2,4% αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν 2,5 εκατομμύρια άδειε. Ε, ενώ θέλουμε να πετύχουμε 700 εκατομμύρια, πολύ, μεγαλύτερους, ε, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε το πλεόνασμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο trading scheme. Αν δεν μειώσουμε το πλεόνασμα, τι κάνουμε. Ε, κάποια στιγμή αργότερα ε, θα έχουμε και πάλι πάρα πάρα πολλές allowances. Γι' αυτό ε, έχει επιτυχία το σύστημα. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές και όταν γνωρίζουμε πόσο επιτυχής την αυτή η διαδικασία βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόκληση. Πρέπει να μην έχουμε υπερπροσφορά allowances και για να πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε πώς θα μπορέσουμε να αποσύρουμε αυτά τα επιπλέον allowances. Το, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ και βοήθησε ιδιαίτερα ο συνάδελφο να το πετύχουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να, συμπληρώσουμε το MSR. Θα υπάρξουν και επιπλέον ε, πλεονάσματα, allowances, και πρέπει να γίνουν απάντητες προσαρμογές. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ δίνω έμφαση στην έκθεση αυτή να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο να το κάνει αυτό. Επιπλέον, όταν εξετάζουμε την προσέγγιση των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά την, την μικρότερη περιοχή τη άνθρακα, την μικρότερη χρήση άνθρακα, ε, δεν είναι ίδια. Ε, δεν πρέπει να ακολουθούμε τον πιο αργό, έτσι δεν πρέπει ο πιο αργό να δίνει το ρυθμό. Ε, εάν δούμε, παραδείγματο χάρη, ποια είναι η ατζέντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Έω το 2025 θέλουμε όλη η ηλεκτρική ενέργεια να έχει χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Για όσου λένε ότι αυτό είναι θελοντικό και δεν πρόκειται να συμβεί, η κάθε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή και έχουν πει ότι πρέπει να έχουν μια φιλόδοξη συμμαχία, πραγματικά θα ντραπούν αν δεν, ε, δεν, θα, αν δεν το πετύχουν αυτό και θα υπάρξει και πίεση από, την κοινή γνώμη. Πρέπει η δέσμευση κάποιου σε ένα χαρτί να μην αρκεί. Θα πρέπει κάποιος μετά να τηρεί τη δέσμευση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αποσυρθούν αυτές οι allowances έγκαιρα ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το πλεόνασμα. Προσπάθησα να αναφερθώ και στα Ηνωμένα Έθνη ε, και στη Συμφωνία του, του Παρισιού αυτή η ανάληψη υποχρεώσεων αφορά το σύνολο και πρέπει να αξιολογήσουμε που βρισκόμαστε. Ιδάλλως το 2023 αντί να αρχίζουμε θα τελειώνουμε. Ε, κάποιοι λένε ότι αν ξεκινήσουμε το 2023 θα πάμε πέρα από το 2030. Αυτό θα γίνει μόνο αν το αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό. Αν ξεκινήσουμε την προπαρασκευή τώρα για το stock taking δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, έτσι ώστε το 2023 θα έχουμε την ε, ε, γενικότερη εικόνα στις χώρες των ΗΠΑ να μην έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Από εκεί και πέρα, και βεβαίως εγώ θα χτεχθώ οποιαδήποτε τροπολογία θεωρείτε εσείς λογική, ε, αναγνωρίζω ότι ε, ε δεν μπορώ βεβαίως να πετύχω όλα αυτά τα οποία θα ήθελα να κάνω μόνος μου. Χρειάζομαι υποστήριξη γι' αυτό, για το κάθε ένα από τα ζητήματα έψαξα τη συνένεση, το συμβιβασμό. Ε, εγώ υποστηρίζω αυτή την έκθεση παρά τις κριτικές, ε, διότι πιστεύω ότι εκεί θα οδηγηθούμε, πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και, και θα, πετύχουμε, θα πετύχει πιστεύω αυτήν την πραγματική αλλαγή εκπομπών που χρειάζεται. Εάν επικεντρωθούμε μόνο στην προσαρμογή ε, ε στην εφαρμογή της μείωσης ε, θα, δεν θα τα πετύχουμε. Το θέμα, το θέμα είναι να φτάσουμε στο στόχο μας, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Συμφωνήσαμε, υπογράψαμε στο Παρίσι. Τώρα θα πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο θα φτάσουμε στο στόχο μας. Όταν πάω από την εκλογική περιφέρεια της Σκωτία στο Στρασβούργο, μπορεί να ακολουθήσω πολλές και διάφορες οδού, αλλά όλες στο Στρασβούργο οδηγούν. Το βασικό είναι να φτάσω στο Στρασβούργο κάθε μήνα. Ξέρουμε πού πάμε. Το θέμα είναι πως θα φτάσουμε εκεί ίσως και με χαμηλή ε, εκπομπή άνθρακα, ακόμα καλύτερα. Κάποια σχόλια ακόμα. Το Ταμείο Καινοτομία θα είναι κρίσιμη σημασία. Ε, ε, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω κονδύλια εκεί. Η καινοτομία είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μειώσουμε το κόστος. Ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει καινοτομία ε, από τη βιομηχανία. Δεν χρειάζεται καν κάποιο ταμείο καινοτομία. Η βιομηχανία εξορισμού από τη φύση τη ε, θα αναστήσει την καινοτομία. Ορισμένε φορέ χρειάζονται όμω κάποια χρήματα για να μπορέσουν αυτέ οι πρώτε ιδέε να αναπτυχθούν. Και ένα τέτοιο ταμείο ε, καινοτομία πρέπει να το κάνει. Πρέπει να είναι πιο δυναμικά τα κονδύλια που διατίθενται. Θα πρέπει ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην αποφελθεί μία ή μία ή άλλη εταιρεία. Μόνο θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα επικεντρωθούμε στο να παρατηρούμε έγκαιρα και όχι καθυστερημένα. Θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι πρέπει να περάσουμε από τους 25 στους 50.000 τόνους, ε, διότι έτσι ε, πολύ μεγάλοι εργοδότες θα βρεθούν εκτός. Εάν το κάνουμε αυτό θα μειωθεί και η γραφειοκρατία. Θα ήθελα επίσης να φύγει το micromeasurements διότι δεν θέλαμε εμεί να καλύψουμε τι επιχεί, τη ε, τα νοσοκομεία ή τις, ε, ε, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Το να του βάλουμε λοιπόν αυτού στο σύστημα δεν έχει νόημα. Η συνεισφορά του στην αλλαγή του κλίματο είναι απειροελάχιστη. Μπορούν να βρεθούν εκτό λοιπόν του συστήματο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν τα συστήματα αυτά έγκαιρα μέσω εθνικών κανονισμών και εθνικών προσεγγίσεων. Αυτό θα καταστήσει το σύστημα πιο διαχειρίσιμο και λιγότερο γραφειοκρατικό. Κάτι τελευταίο. Η κυβέρνησή μου ήθελε μια προσέγγιση ε, σε δύο ταχύτητες, διάφορες ταχύτητες. Ε, νομίζω ότι πρέπει όμως να, να μην συμφωνούμε παρά με την κυβέρνησή μας. Ε, και εγώ αυτό έκανα, βρήκα ένα καλύτερο τρόπο να το κάνω αυτό. Πρέπει αυτή την tiered approach να την εξετάσουμε. Υπάρχει αυτός ο, ο παράγοντας διόρθωσης, ο διατομιακός, αλλά είναι πραγματικά προβληματικό αυτό για κάποιον ο οποίος ε, έχει 100% allowances. Είναι άδικο λοιπόν να πάρουμε το πιο αποτελεσματικό και να τον ε, ε, τιμωρήσουμε ουσιαστικά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να το, αντιμετωπίσουμε αυτό εξετάζοντας αυτό το tiered system. Πιστεύω ότι λειτουργεί. Μία από τις πολιτικές ομάδες μας φάνηκε φιλόδοξη και πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτός ο παράγοντας διόρθωσης δεν είναι το κατάλληλος. Ε, ελπίζω να μην χρειαστεί ε, να ξεκινήσει η διαδικασία. Λοιπόν, δεν σας κουράσω άλλο. Πολλά έχω να σας πω. Έχω πολλές ιδέες. Να πω απλώς ότι πραγματικά χάρηκα που συνεργάστηκα με τους κοινότητες, συζητητές. Ήταν ανοιχτή, ε, ήταν συνεργάσιμη πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μέρο τη διαδρομή. Θα βρούμε τι κατάλληλε συμβαστικέ λύσει, θα εξασφαλίσουμε ότι η φιλοδοξία που έχουμε ε, θα φέρει επιτυχία. Ε, πιστεύουμε ότι η φιλοδοξία των συμφωνία του Παρισιού μας οδηγεί προς νέους προορισμούς. Θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα, θα βρεθεί συνένεση, θα μπορέσουν να προχωρήσουν τροπολογίες. Είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε και είναι και ο κατάλληλος τρόπος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους κοιόδες συγκητές και αναμένω με ανυπομονησία ε, τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Duncan. Ευχαριστούμε κύριε Duncan. Πρωτού αρχίσουμε το συνηθι γύρω ερωτήσεων, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Ε, αναφέρομαι στην πρόσθετη δήλωση που κάνατε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε πεπισμένοι εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι και μετά την 23η Ιουνίου θα εξακολουθείτε εσείς να είστε ο εισηγητής μας. Αυτό ελπίζουμε. Και θέλουμε να συνεχίσετε τη δουλειά που ξεκινήσατε. Ας αρχίσουμε τώρα. Ήβο, Ελκ. Ευχαριστώ. Και εγώ αυτό θέλω να τονίσω, την ίδια παρατήρηση ήθελα να κάνω. Διάβαζα στον τύπο χτες τι θα γίνει αν συμβεί ε, το απευκταίο. Εμείς ε, υπολογίζουμε σε εσά, ε, βασιζόμαστε σε εσά, θέλουμε να παραμείνετε εδώ, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι εξαιρετική η βάση ε, των μελλοντικών μας εργασιών και διαπραγματεύσεων χάρη στις ε, πολυέρθμες προτάσεις που καταθέσατε. Είμαστε αισιόδοξοι πάντως. Παραμένουμε αισιόδοξοι για την κατάσταση μετά την 23η Ιουνίου. Για την Ενεργειακή Ένωση ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε και επιτρέψτε μου Πρόεδρε να κάνω και μια παρατήρηση διότι είμαι κάπως πιο αισιόδοξο ε, σε σχέση με τις ε, δυνατότητες εφαρμογής. Ο κύριος Σεύκοβιτς θα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό για την Ενεργειακή Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω θα συνεργαστεί με τον διότι το Ηνωμένο είναι στην καρδιά της, Ευρωπα... της Ενεργειακής Ένωσης, οπότε δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος. Πολλά ε, θετικά στοιχεία λοιπόν στην έκθεση Duncan αναφερθήκατε στο Παρίσι και δικαίως. Φυσικά θέλουμε να τηρούμε τις ε, διεθνείς μας υποχρεώσεις και να ε, τηρήσουμε το μείον 40% για το 2030 και για το ε, μείον 30%. Ε, Αναφερθήκατε και στο περίφημο split, δηλαδή το διαχωρισμό ανάμεσα στις άδειε που δημοπρατούνται αφενός και αφετέρου στις δωρεάν άδειες. Ε, χαίρομαι που δεν κλείνεται αυτό, αυτή την πόρτα. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες εξάλλου για να αρχίσει η συζήτηση για το διαχωρισμό αυτό ανάμεσα στις δημοκρατούμενες άδειες και τις δωρεάν άδειες. Ε, ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την μία και η βιομηχανία από την άλλη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια συζήτηση θα έχουμε πλέον τα πετούμενα στοιχεία στη διάθεσή μας για να δώσουμε και απαντήσεις. Ε, κάτι άλλο στο οποίο δεν εστιάσατε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο ETS, ε, στο σύστημα ε, δικαιωμάτων εκπομπών, αλλά ε, πρόκειται για αλληλένδετα ζητήματα, διότι και στους κλάδους μη ETS, όπως τον κατασκευαστικό και στον τομέα των μεταφορών, χρειαζόμαστε κάποιο περιθώριο ελιγμών. Ε, και αυτό θα το επιτύχουμε χάρη στους τομείς ε, μη ETS. Ε, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το καταφέρουμε αυτό, αλλά πάντως θα καταθέσουμε τροπολογίες, κυρίως για την αεροπορία, ώστε το ε, όριο για την αεροπορία ε, να ε, ευθυγραμμιστεί με τα εσωτερικά όρια, δηλαδή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαρροή άνθρακα. Τους τελευταίους έξι μήνες συζητούμε αυτό το ζήτημα και υπάρχει η tiered approach, όπως μας είπατε, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Αυτή η προσέγγιση σταδιακή που μας προτείνεται μας επιτρέπει ε, τελικά να επιστρέφουμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς αυτό έχουμε καταλήξει. Ίσως βρεθεί μια μέση οδός, αλλά ε, αυτή η ε, η ε, διπλή προσέγγιση ε, που μας προτείνουν οι σοφοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας φαίνεται η καλύτερη λύση. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αναφερθήκατε και στα σημεία σύγκριση. Τα benchmarks είναι ε, ζωτική σημασία για ολόκληρη τη διαδικασία. Αναφερθήκατε στον πραγματικό χρόνο και όχι σε ιστορικά δεδομένα. Ακριβώς συνοψίσατε με ακρίβεια την κατάσταση. Θα καταθέσουμε τροπολογίες ώστε να επικαιροποιηθούν τα benchmarks επί τη βάση πραγματικών επιδόσεων και εξακρίβωση των στοιχείων να προτού αρχίσει η εμπορία των δικαιωμάτων. Αλλά εξάλλου έχετε καταθέσει και εσείς ε, ε, προτάσεις. Θα καταθέσουμε επίσης ε, τροπολογίες για άλλα ζητήματα. Σε σχέση με το auction share για τις δημοκρατήσεις δηλαδή και την τιμή των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να καλύψουμε το επιπρόσθετο κόστος. Ε, δεν είναι η ε, ισότιμη η όρη ανταγωνισμού και θέλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, χρηματοδότηση για την καινοτομία. Επίσης, χέρια σημασίας. Και να προσθέσω και ένα σημείο, Πρόεδρε, εισηγητά, ίσως είναι υπερβολικά λεπτομερείς οι κανόνες και τα κριτήρια και ξεχνούμε ότι πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση, μην ξεμείνουμε και από κονδύλια για τους μικροεκπομπούς, micro emitters, συμφωνούμε και πώς ε, ε, συνδέεται ε, το ETS με την ενεργειακή αποδοτικότητα, με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή κάποιοι εμπλεκόμενοι φορείς μιλάνε για λεπικάλυψη. Όχι, είναι διάδραση των διαφόρων πολιτικών όπως με την πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει ολιστικά να προσεγγίζουμε το ζήτημα. Αυτό που προτείνεται μας βρίσκει σύμφωνος ότι είναι απαραίτητο να ε, κάνουμε έναν απολογισμό ε, του συνδυασμού των πολιτικών της Ένωσης. Ευχαριστούμε. Welchen Namen der Bericht in Zukunft tragen wird, ich würde mir wünschen, dass Sie Ihnen danken, weiterhin der Berichterstatter ist, aber es wie im Leben das normal so ist, ist es eine Wahl. Insofern äh,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 Für Sie ist es για τη Σκιώδη ήταν σημαντικό να υποβληθούν τροπολογίες σε σχέση με το επίπεδο των φιλοδοξιών και παράλληλα να γίνει πιο προβλέψιμη η νομοθεσία για τη βιομηχανία για όλους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλους τους δρόντες. Πρέπει να υπάρχει μια λογική ισορροπία. Το κύριο πρόβλημα του υφιστάμενου συστήματος είναι ότι έχουμε υπερβολικό ρυθμό πιστοποιητικών στην αγορά. Πρέπει να ασχοληθούμε διεξοδικά με το ζήτημα και είναι πολύ πιθανό αυτό να πονέσει. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε ταυτόχρονα για τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε στην πρώτη κοινοβουλευτική περίοδο αυτό ήταν πολύ ακραίο να αποφύγουμε Α, αποφύγουμε τα πρόσμενα κέρδη. Πρέπει επίση να βρίσουμε για τη μεταβατική περίοδο τη αποδέσμευση από τον άνθρωπο σε εκείνε τι περιφερειέ που χρειάζονται υποστήριξη και πρέπει να σκεφτούμε του ανθρώπου που εργάζονται και ζουν σε τέτοιε περιφερειέ, επειδή εκεί αυτοί βλέπουν την Ευρώπη. Κύρια σημεία για την σοσιαλδημοκρατική πολιτική ομάδα είναι το επίπεδο. Πρέπει να προσαρμόσουμε τον γραμμικό συντελεστή. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει 2,2%. Εμείς προτιμούμε 2,4%. Πρέπει, δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να επιτρέψουμε νέα πιστοποιητικά. Αυτό σημαίνει πως τα πιστοποιητικά πρέπει να διαγραφούν από τα αποθεματικά στο τέλος της ισχύω τους και πιστοποιητικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να διαγραφούνται επίσης. Όσον αφορά τη διαρροή του άνθρακα, χαιρετίζουμε τον περιορισμό στο 34%. Απομένουν 57% για τη δημοπράτηση. Εμείς ως πολιτική ομάδα συμφιλωνόμαστε με την πρόταση αυτή αλλά θέλουμε και το τονίζω αυτό η δωρεάν κατανομή να αποτελέσει μια εξαίρεση στο σύστημα. Σημαντικό είναι για μας σημαντική είναι η ευελιξία κατανομής στο σύστημα και να έχουμε ένα περιθώριο απρικούς μεγέθους. Η πρόταση της Κομισιόν επικυρωποιεί τους δείκτες αναφοράς μια πιο στοχευμένη προσέγγιση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει καλύτερα τους τομείς μεταξύ τους και να καταστεί όλη η διαδικασία πιο δίκαιη. Συμφωνούμε καταρχήν με τον εισηγητή. Ωστόσο, εμείς θα προσεγγίζαμε το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε πως δεν θα έχουμε πίσω πόρτες ανοιχτές. Όσον αφορά τη στοχευμένη προσέγγιση από την αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν είναι μια καλή βάση, η οποία πρέπει ωστόσο να εκτεπτυνθεί ακόμα. Το μοντέλο, ο εισηγητής ακολούθησε το γαλλικό και το βρετανικό μοντέλο. Εμείς ως S&D είμαστε της άποψης ότι με την εκτέπτυνση η Κομισιόν δημιουργεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι στη συζήτηση δεν θα έχουμε τον κίνδυνο, οι συνήθεις ύποπτοι να έρθουν, πως πρώτα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου και αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, αντί ενός διτού μοντέλου της πρότασης της Κομισιόν, κατά την οποία η βιομηχανία παίρνει είτε 30 είτε 100% δωρεάν κατανομές, θα μπορούσε να ακολουθηθεί ένα, μια διαφορετική κατανομή. Δωρεάν κατανομή δεν θα πρέπει να δίνεται σε τομείς που δεν βρίσκονται στην, στον κατάλογο διαρροής άνθρακα. Η κατανομή πρέπει να γίνεται ανά 10 χρόνια για τον καλύτερο σχεδιασμό, αλλά συχνή επικαιροποίηση των δεδομένων παραγωγή και μια καλύτερη βάση δεδομένων χρειαζόμαστε ανά 5 έτη και όχι ανά 10. Σημαντικό είναι επίσης να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε την καλύτερη επίδοση και να δώσουμε κίνητρα. Εμείς ως SED θέλουμε περαιτέρω κλιματικά μέτρα. Αυτό το είπαμε ήδη στην πρώτη συζήτηση για τη συμπερίληψη των εναέριων μεταφορών. Στην κλιματική, η κλιματική αλλαγή θα, θα κοστίσει πολλά χρήματα. Επίσης η προσαρμογή ως προς το κλίμα. Και πιστεύω, όπως και η πολιτική ομάδα, πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα τα χρήματα αυτά όσον αφορά την αποζημίωση για έμεσα έξοδα. Εδώ θέλουμε να κινήσουμε ένα ευρωπαϊκό ε, σύστημα για να αποφευθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Όσον αφορά τα ταμεία, αφενός έχουμε το Ταμείο Καινοτομίας, αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί κατά την απόψή μας, έτσι ώστε να υποστηρίξει την βιομηχανία κατά την υλοποίηση. Ταυτόχρονα θέλουμε σαφή κριτήρια για την επιλογή. Για το Ταμείο Εξυγχρονισμού θέλουμε να διασφαλίσουμε πως τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται εκεί να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θέλουμε διαφάνεια. Δεν θέλουμε να δρομολογηθούν πράγματα για τα οποία μπορεί να διερωτηθεί κανείς εκ των υστέρων εάν αυτό είναι εξυγχρονισμός. Δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σημαντική είναι επίσης η θέσπιση ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και εδώ θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τους τομείς όπου παρουσιάζεται κοινωνική σκληρότητα. Το Ταμείο αυτό θα είναι συμπληρωματικό στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να βοηθήσει σε τομείς όπου ίσως οι άνθρωποι λόγω της μεταβολής της, της κοινωνίας συγγνώμη, σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα υποστούν συνέπειες. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ε, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία για τα οποία συζητούμε συνέχεια, με τα οποία ασχοληθήκαμε και στην κλιματική σύνοδο. Είναι η πλοία και οι εναέριες μεταφορές. Κατά την άποψή μου και οι δύο τομείς πρέπει να ρυθμιστούν σε διεθνές επίπεδο γνωρίζετε ότι πολλές φορές η πρόοδος επιτυχάνεται με ρυθμό σαλιγκαριού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το σαλιγκάρι πρέπει να τρέξει λίγο γρηγορότερα. Θέλουμε να υπάρξει ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο. Αλλά εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και για τους δύο τομείς πώς μπορούν να συμπεριληφθούν. Επειδή δεν αποτελούν παρά ένα μικρό τμήμα αυτών που προκαλούν εκπομπές, είναι 8%, αλλά αναπτύσσονται πολύ έντονα. Γι' αυτό και προτεραιότητα έχει μια διεθνή ρύθμιση. Αν, αλλά αν δεν μπορέσουμε να την επιτύχουμε, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον μπορούμε να ελέγξουμε το όλο ζήτημα. Αυτά από την πλευρά μου για την σκιώδη συγκήτρια μας, Γιούτε Κούτελαντ και την πολιτική μας ομάδα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει εδώ κάποιο από του φιλελεύθερους, από την ΚΟΕ, από τους πράσινους, από το Γεφτιντή είναι εδώ και ο συζητητής. Η κυρία Τορνάνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντάνκαν για αυτό το μακρύ και κουραστικό έργο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που πέτρεψε ε, ανταλλαγή απόψεων με τον οικονομικό κόσμο, τον μηχανικό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών. Συμμεριζόμαστε μεγάλο μέρο των προτάσεων του εισηγητή. Όμω, θέλω να τονίσω και τι διαφορέ μα. Ε, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση τη σταδιακή και το θέμα του άνθρακα έχουν πολλέ επιφυλάξει και η πρόταση τη Κομισιόν δεν ήταν ικανοποιητική. Μπορεί κάποιοι μεγάλοι μολυντέ και εξαγωγείς να παραμένουν ε, σε προτιμησιακό καθεστώς ε, άλλοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που έχουν πολύ σημαντική προσθέμενη αξία στην παραγωγή τους δεν θα προστατεύονται πια. Και αυτό αποτελεί διαστρέβλωση του ανταγωνισμού. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την έκθεση. Οι κλιματικοί στόχοι δεν πρέπει να καταστρέψουν τη βιομηχανία μας. Και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και αυτή η προσέγγιση σταδιακή, ουσιαστικά μας οδηγεί στο να αυτοτραυματιζόμαστε. Ε, επίσης διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι και οι απαιτήσει οι, περιβαλλοντικοί, αφορούν το σύνολο τη οικονομία μα. Στο άρθρο 1, 4, DB, που έρχεστε να τροποποιήσετε όμω, μιλάτε για διάδραση με τι περιβαλλοντικέ και ενεργειακέ πολιτικέ. Πρέπει όμω αυτό το συντονισμό να τον επεκτείνουμε, να καλύπτουμε και τι μεταφορέ που είναι σημαντική ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Επίση, το σύστημα, το πρώτο θέμα των δωρεάν ε, allowances πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια μια ευρύτερη ε, προσέγγιση. να προστατεύσουμε δηλαδή όλου του παράγοντε και όλα τα στάδια τη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ε, αυτόν τον τομέα τον εξετάζουμε υπό το πρίσμα τη ε, αποσύνδεση τη αγορά από τις, βιομηχανίε δικτύου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Λίζε έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ επίσης τον Ιαν Ντάνκαν. Ζητώ συγγνώμη που άργησα λίγο. Δεν μπόρεσα να φανταστώ ποσά προχωρούσαμε τόσο γρήγορα. Παρά τα αυτά, είναι κρίμα που οι σκιώδεις των άλλων πολιτικών ομάδων δεν είναι εδώ. Ίσως μπορεί κάποιος να τους πάρει τηλέφωνο, να δούμε που είναι. Επειδή πρέπει να έχουμε μια εκτενή συζήτηση. Εμείς από το ΕΛΚ Θέλουμε μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική, αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε πως δεν θα υπάρξει διαρροή άνθρακα. Πως δηλαδή δεν θα εξαναγκαστούν επιχειρήσεις να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές όπου οι κανόνες είναι λιγότεροι αυστηροί. Πιστεύουμε πως με μονομένοι τομείς έχουν πρόβλημα με την πρόταση της Κομισιόν, η οποία δεν είναι κακή, αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Το πιο σημαντικό είναι πως χρειαζόμαστε περισσότερο, περισσότερες δωρεάν κατανομές για επιμέρους τομείς οι οποίοι σε ευρωτική περίπτωση διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Για να λύσουμε το πρόβλημα μπορούμε να μειώσουμε λίγο το μερίδιο της δημοπράτησης. Πιστεύω πως τα κράτη-μέλη μπορούν να το αντέξουν αυτό, επειδή αν φύγουν επιχειρήσεις έχουν λιγότερα φορολογικά έσοδα και αυτό δεν είναι προς συμφέρον των Υπουργών Οικονομικών και δεν είμαι τόσο σίγουρος πως αν περιορίζαμε λίγο το μερίδιο της δημοπράτησης θα υπήρχαν λιγότερα έσοδα για τα εκάστοτε Υπουργεία Οικονομικών. Επειδή με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται έλλειψη διαθεσιμότητας, οπότε και πάλι αυξάνεται η τιμή. Το 10% των καλύτερων πρέπει να παίρνουν 100% δωρεάν κατανομή. Το δεύτερο θέμα που έχουμε είναι οι εναέριε μεταφορές, είτε θέλουμε είτε όχι, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε για τις εναερίες μεταφορές με τις άλλες βιομηχανίες. Και εκεί θα δούμε πως έχουμε μόνο ένα στόχο μείωσης κατά 10% ενώ στο χάλιβα, στο τσιμέντο κτλ. Έχουμε ένα στόχο Τη τάξη του 43%. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω σε κανέναν χαλιβουργό που μάχεται για τη θέση εργασία του, ότι πρέπει να έχει την τετραπλάσια μείωση από αυτήν των εναέριων μεταφορών. Στι εναέριε μεταφορέ έχουμε διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίο ωστόσο δεν είναι οξύτερο από ό,τι στη χαλιβουργία. Το τρίτο στοιχείο που πιστεύω ότι έχει κάποιο περισσότερο περιθώριο είναι η σχέση μεταξύ ETS και effort sharing. Γνωρίζω ότι σας αντιδράσουν τα κράτη-μέλη, αλλά η κατάσταση είναι σαφής. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Γιούγκερ, είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως χρειαζόμαστε ένα στόχο τουλάχιστον της τάξης του 30%. Τώρα το έχουμε προσδιορίσει στο 27%. Υπάρχει μια αίτηση του ΕΛΚ για την ψηφοφορία της Πέμπτης, για την έκθεση του Μάρκος Λίπα, όπου λέμε τουλάχιστον 30%. Μπορούμε να πούμε δηλαδή πως η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι υπέρ της αύξησης του στόχου ως προς τις εκπομπές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά τουλάχιστον στα 30%. Εάν αυτό είναι έτσι, τότε θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση στον τομέα του εφοσέριν, στον τομέα των κτηρίων. Και εκεί μπορούμε να δώσουμε κάποια περιθώρια ίσως στη βιομηχανία, με το να είμαστε λίγο πιο, λίγο πιο ελαστικοί στο ETS. Τα κράτη-μέλη θέλουν λιγότερη ελαστικότητα. Εμείς θέλουμε στο FOSR να επισπεύσουμε τα πράγματα και να θυμίσουμε την ευθύνη που έχουμε για την προστασία του κλίματος. Εάν διασφαλίσουμε πως οι βιομηχανίες που απειλούνται από διαρροή άνθρακα τύχουν καλύτερη μεταχείριση. Εάν στα 10% τους καλύτερους δώσουμε όντως 100% δωρεάν κατανομές, τότε από την προσωπική μου απόψη μπορούμε να μιλήσουμε επίσης για ένα φιλόδοξο σχέδιο. Τώρα κατά πόσο θα αυξήσουμε τον γραμμικό συντελεστή η δική μου πολιτική ομάδα είναι σκεπτική ως προς αυτό, αλλά τίθεται επίσης το ερώτημα πότε θα αρχίσουμε με, τον, με τη νέα πορεία μείωσης. Πότε θα πάμε από το 1,7 στα 2,2. Από την άποψή μου πιστεύω πως πρέπει να το κάνουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε υπερεκπληρώσει τον στόχο του 2020, αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί. Κατά την υλοποίηση της πολιτικής μας για το 2030. Θα φέρω ένα παράδειγμα από την ιατρική που μου οδηγήθηκε χτες ένας ειδήμονας. Όταν πάμε στον γιατρό, ας φανταστούμε πως είμαστε υπέρβαροι και ο γιατρός μας λέει πως πρέπει να χάσουμε 30 κιλά, οπωσδήποτε. Στα επόμενα δύο χρόνια, αλλιώς θα, πάρετε, πάθετε διαβήτη, εγκεφαλικά και άλλες σοβαρές νόσους. Και όταν χάσουμε μετά το πρώτο έτος 20 κιλά, τότε θα ήταν λάθος στρατηγική να τρώμε κάθε μέρα μία τούρτα με σαντιγή. Καλύτερα θα ήταν να συνεχίσουμε έτσι. Έτσι είναι και η προστασία του κλίματος. Όταν έχουμε πάρει μια καλή πορεία δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία που όπως την αρχίσουμε. Μια παρατήρηση για το τέλος. Το ELK είναι κατά το TFT approach. Ωστόσο δεν έχω ολοκληρώσει τις σκέψεις μου για τις επιχειρήσεις που είναι οριακά που δεν παίρνουν το 100% της κομισιόν, που δεν ανήκουν στην κατηγορία 1. Πιστεύω πως τουλάχιστον θα μπορούσε να εξετάσει κανείς κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Γιατί χρειαζόμαστε κατηγορίες. Γιατί μπορούμε να πούμε ή 100% δωρεάν ή 30% και μετά τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε αντί για κατηγορίες να έχουμε μια καμπύλη έτσι ώστε ο καθένα ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει να υποστεί διαρροή άνθρακα, να κατανεμηθεί και να λάβει μια δωρεάν κατανομή. Δηλαδή όχι 100 ή 30% ή 100 ή 80% αλλά ο καθένα να έχει αυτό που αξίζει, 85-55%. Αυτός ίσως είναι και ένας τρόπος για να μειωθεί λίγο ο λομπισμός Και η κατηγοριοποίηση αυτή έχει συνέπειες αξίας δισεκατομμυρίων. Με μια καμπύλη οι συνέπειες ίσως ήταν πιο ομαλές. Επίσης, Εμεί από το ΕΛΚ θέλουμε να εξεταστεί κατά πόσον οι όντω καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να επιβραβευθούν λίγο καλύτερα. Επειδή στα αυτοκίνητα έχουμε τα super credits. Όποιος είναι πάρα πολύ καλό, όποιο υπερεκπληρώνει το στόχο, παίρνει μια πίστοση θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς κατά πόσον οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν μόνο στο 10% των καλύτερων, αλλά αυτές που είναι οι καλύτερες απολύτως, που υπερεκπληρώνουν τους στόχους, κατά πόσον θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερα δωρεάν δικαιώματα για να έχουν κάποιο κίνητρο, όχι δηλαδή μόνο να μην τιμωρούνται, αλλά να κερδίζουν από την καινοτομία τους, από την προστασία του κλίματος. Όσον αφορά το Ταμείο Εξυγχρονισμού, υποστηρίζω αυτό που είπε ο Ματίας Γκρότε, Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς να είναι όντως εξυγχρονισμός να μπούμε στον δρόμο της μακροπρόθεσμης προστασίας του κλίματος. Εάν τα καταφέρουμε, εγώ προσωπικά θα ήμουν της άποψης το Ταμείο Εξυγχρονισμού, ότι το Ταμείο Εξυγχρονισμού θα μπορούσε να λάβει περισσότερα, περισσότερους πόρους. Και υπάρχει μια λύση στο άρθρο 10C, έχει προταθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας να υπάρχει επίσης δωρεάν κατανομή. Ίσως ήταν καλύτερα να πούμε πως θα αυξήσουμε το Ταμείο Εξυγχρονισμού έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ως προς την καινοτομία, η δωρεάν κατανομή θα μπορούσε ίσως να διατηρήσει φυστάμενες δομές για υπερβολικό χρονικό διάστημα. Και ως προς το τελευταίο σημείο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Γκρότε, τα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να ξοδεύονται με στοχευμένο τρόπο. Μιλάμε για ένα εργαλείο που είναι για την προστασία του κλίματος και όχι για την διάσταση του προϋπολογισμών. Αυτό πρέπει να το διατυπώσουμε πιο σαφώς από ότι αναφέρεται στο σχέδιο της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πότς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτή είναι μια νέα απόπειρα να διορθώσουμε το σύστημα αυτό. Ελπίζω σε μια πενταετία να μην είμαστε πάλι εδώ και να συζητάμε και πάλι πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το ισχυρό σύστημα, εάν ναι. Εάν ε, τα καταφέρουμε, ελπίζω να γίνουν ε, ε, αποφασιστικές σημασίες αλλαγές. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για το Linear Reduction Factor, το γραμμικό συντελεστή μείωσης. Έχει κατατεθεί η πρόταση αναθεώρησής του. Πολύ καλό αυτό. Αυτό όμως πραγματικά θέλουμε σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Τι χρειαζόμαστε γι' αυτό, χαμηλό γραμμικό συντελεστή, ε, αλλά το επιδιώκουμε αυτό μόνο και μόνο για να μπορέσει να εγκριθεί, ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν υποστηρίζει μακροχρόνια μείωση ε, των εκπομπών άνθρακα. 2,4 αντί για 2,2 λοιπόν και ας προτείνουμε νέα αναθεώρηση μετά από 6 χρόνια. Ε, λένε κάποιοι. Μα γιατί να μην το κάνουμε κατευθείαν, ε, αφού, αφού επιδιώκουμε την σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στις αγορές. Ε, δηλαδή θα υιοθετήσουμε προσωρινά ένα στελεστή και ο οποίος θα αναθεωρηθεί μετά από έξι χρόνια. Δεν είναι σωστή ε, λύση για τις δημοπρατήσεις. Ε, 57% είναι το ποσοστό που, που προτείνεται. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς πώς κατέληξε αυτό το ποσοστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω δει και υπολογισμούς που οδηγούν στο 59% ή σε άλλους που μου καταλήγουν στο 52%. Ε, απευθύνω το ερώτημα στην Επιτροπή. Γιατί λοιπόν καταλήξατε σε αυτό το ποσοστό. Επίσης, δεν θα πρέπει και εδώ να προβλέψουμε μια ε, αναθεώρηση ενδιάμεση για το benchmarking, της ε, τις τιμές σύγκρισης, ε, θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και το CCS, διότι για κάποια κράτη-μέλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι υπερβολικά ε, ακριβό το σύστημα. Δεν, ε, ξέρουμε ότι δεν ε, αναπτύσσονται ομοιόμορφα όλες οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήστε που δεν συντρέχουν και οι γεωλογικές προϋποθέσεις, ούτως ώστε να έχουν τέτοιες υποδομές δέσμευσης άνθρακα. Επίση, γιατί δεν αναφερόμαστε στη δασοκομεία. Η δυνατότητα δέσμευση του άνθρακα στα δάση είναι μια ε, πολύ ε, ευνοϊκότερη, φθηνότερη και μακροπρόθεσμη λύση. Για το αποθεματικό της αγοράς, το αποθεματικό ασφαλεία. ναι, είναι ένα εργαλείο, όμως μην ξεχνάμε ότι ε, είναι προϊόν μια εξαιρετικά πολύπλοκη πολιτικής συμφωνία και αν αποκλίνουμε από τη συμφωνία για το αποθεματικό, νομίζω θα είναι ε, δυσμενείς οι επιπτώσεις. Το Ταμείο για την Καινοτομία, για να περάσω σε κάτι άλλο, θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να μην λαμβάνεται υπόψη ε, και ο παράγοντας της γεωγραφικής ισορροπίας, όπως δηλαδή είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν το αποφασίσουμε... Και αν δούμε τι έχει συμβεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φυγόκεντρες τάσεις ε, κάποιων κρατών μελών, Αναφέρθηκε ο κύριο Ντάκαν εξάλλου σε αυτό στην αρχή τη παρέμβασή του. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη τη παρελθού εμπειρία, δεν κρίνω ότι η απάλληψη του παράγοντα τη γεωγραφική ισορροπία είναι μια πολύ καλή ιδέα και με ξαφνιάζει που την επέβαλε αυτή την ιδέα ο κύριο Ντάκαν εξάλλου. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάνκαν που εργάστηκε σκληρά επ' αυτού του σχέδιου έκθεσης για το ETS. Και το αποτέλεσμα το δέχομαι με συγκρατημένη ικανοποίηση. Χαίρομαι που παραμένει αυτός ο συντελεστής ε, για την μείωση των εκπομπών που εγκρίθηκε το 2014 ε, και που μειώνεται σταδιακά υπό αυτή τη μορφή σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές οι απαιτήσει αποτελούν σημαντική πρόκληση για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει αύξηση, περαιτέρω αύξηση. Εδώ γίνεται αναφορά στην δυνατότητα αύξηση του τελεστή μετά το 2023. Μετά δηλαδή από την αξιολόγηση όλων των συμβαλωμένων μερών στη Συμφωνία του, του Παρισιού. Αυτό αιτιολογείται μόνο εφόσον όλες οι χώρες που εκπέμπουν ε, διοξείδιο του άνθρακα συμφωνήσουν. Ιδάλως ε, υπονομεύουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Το γεγονός και μόνο ότι η Συμφωνία του Παρισιού υπογράφηκε ε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι συμβαλόμενοι θα κάνουν κάτι ενεργά για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι ο εισηγητής αναφέρει το γεγονός ότι πρέπει να προστατέψουμε την βιομηχανία μας στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό νομίζω ε, ότι τονίζει ε, γενικότερη απειλή για την οικονομία από το carbon leakage ο εισηγητής. Επίσης πρέπει να υποστηριχθούν ε, τα εργοστάσια ε, παραγωγής. Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου μπορεί να υπάρξει βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλη που δεν μπορεί να συμβεί αυτό, όπως στον τομέα του χάλιβα, όπου υπάρχει σημαντική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Ε, αυτό συμβαίνει και στον τομέα των λοιπασμάτων, παραδείγματος χάρη. Ε, χαίρομαι που συμφωνεί ο εισηγητή να έχουμε έναν πιο εύκολο τρόπο για να ένα πιο απλό τρόπο για να μπορέσει κάποιο να σέβεται το συντελεστή αυτό. Το... Θα ήταν βέβαια καλύτερο αυτοί οι δείκτες, αυτοί οι να εξεταστούν πιο ρεαλιστικά. Οι άλλες προτάσεις που αφορούν άλλου τομεί που έχουν χτυπηθεί από την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης ε, όλα αυτά αποτελούν μια καλή βάση συζήτησης, ε, παρότι δεν είμαι βέβαια ενθουσιώδης. Ε, η δυνατότητα διαφοροποίησης του αριθμού των, ε, των allowances ανάλογα με τη δυνατότητα carbon leakage που έχει ο κάθε κλάδος, καθώς και ο, μηχανο, ο μηχανισμός ευελιξίας που θα μας επιτρέψει να χορηγήσουμε επιπλέον ε, πόρους σε μία σε έναν κλάδο βιομηχανικό, αυτό το βρίσκω, αυτό το βρίσκω κάπως προβληματικά. Ο εισηγητής πάντως έχει πάρει μια πολύ σωστή στάση σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αντιστάθμισης. Ε, η λύση που προτείνεται για να, καλυφθεί, να καλυφθούν ε, τα κράτη-μέλη που έχουν ΑΕΠ κάτω από 60% του ευρωπαϊκού Μεσόρου και που έχουν πληγεί από την πολιτική, την παραγωγική πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, ε, είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το κόστος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Βεβαίως συμφωνώ ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή δηλαδή προτείνει ο εισηγητής. Ε, αντίθετα με τις προηγούμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντάνκαν πρότεινε να μειώσουμε σημαντικά τη διαχείριση των μηχανισμών σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση. Πρότεινε πολλές οντότητες να έχουν ένα περιορισμένο ρόλο εδώ. Καλωσορίζω επίσης την πρότασή του σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κατοφλίου, σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τα αιτήματα δημοσίων προμηθειών εδώ θα πρέπει να δούμε και το θέμα της μεταβίβασης τεχνολογίας, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Θεωρώ βεβαίως ότι οι διαδικασίες δημοσίων προμηθειών δεν είναι απαραίτητες και πρέπει να αφήσουμε τα επενδυτικά προγράμματα να προχωρήσουν. Συμφωνώ όμως με την ιδέα, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα οικονομικής υποστήριξης στα πλαίσια των μηχανισμών αντιστάθμισης πρέπει να είναι απολύτως διαφανή και βεβαίως ε, να ελέγχονται δημόσια. Επίσης ε, χαίρομαι υπάρχουν προτάσεις για την διοικητική απλοποίηση και τη δυνατότητα να εξαιρέσουμε τις πιο μικρές εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι ο κ. Ντάκαν προτείνει να ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση που μας επιτρέπει να δώσουμε έτσι μεγαλύτερο ρεαλισμό σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φλόρενς. Äh, ο συνάδελφος Τάνκαν άρχισε την τοποθέτησή του με την ερώτηση την πέμπτη ναι ή όχι. Και πρέπει να αντιδράσω πάνω σε αυτό. Επειδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είμαι πολύ υπέρ του να παραμείνει εδώ Θέλω πολύ ο κύριος Ντάγκαν να συνεχίσει να εκπονεί την έκθεση. Αλλά όποιος μετά από μια τόσο επίπανη διαδικασία πει όχι, θα γνωρίσει τις συνέπειες εκ μέρους μου. Όποιος πει όχι πρέπει να το δεχτεί. Δεν θέλω να σταματήσω τη συζήτηση, είναι η προσωπική μου άποψη. Μην κατηγορήσετε το ΕΛΚ γι' αυτό, αλλά αν μετά από αυτή την πολύχρονη συζήτηση πείτε όχι, τότε δεν αρκεί να δώσετε την έκθεση στην πολιτική σας ομάδα, αλλά η πολιτική σας ομάδα πρέπει να σκεφτεί κατά πόσο θα παραγγείλει την Παρασκευή το φορτηγό για τα έπιπλα. Αυτή είναι η απόψή μου. Είτε μέσα είτε έξω. Αυτό ήθελα να πω σαφώς. Μη μου πείτε μετά πως δεν έχω τη δυνατότητα να προβώ σε συγκρούσεις. Ναι, μπορώ να μαλώσω, να αρχίσω καυγάδες όσο μεγάλη και αν είναι η ανεκτικότητά μου. Υπάρχουν εσείς τα επιχειρήματα ότι έχει γεννήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν αποφασίσετε, παρακαλώ, μην δώσετε απλά σε άλλους την έκθεση, αλλά παραγγείλετε το φροντιό για τα έπιπλα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον καιρό να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ο κύριος Λάινεν. Ας ελπίσουμε πως το φορτηγό με τα έπιπλα δεν θα χρειαστεί να έρθει. και πώς θα συνεχίσουμε την κοινή πολιτική μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Γι' αυτό και θα ήθελα ο κύριος Ντάνκα να συνεχίσει να εποπτεύει τον φάκελο αυτό. Γνωρίζω πόσο επίπονη ήταν η διαδικασία τους τελευταίους μήνες. Να ακούσει όλους τους ενδιαφερόμενους, να διαμορφώσει μια άποψη. Και πιστεύω πως συμμερίζομαι με όλους τους συναδέλφους την άποψη πως η πολιτική προστασία του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι αξιόπιστη. Το οποίο σημαίνει επίσης πως τα εργαλεία μας πρέπει να είναι αξιόπιστα. Και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων στην τρίτη φάση του δυστυχώς δεν πληρεί τους στόχους του. Ως εκ τούτου η μεταρρύθμιση του είναι απαραίτητη έτσι ώστε το σύστημα αυτό να ενδυναμωθεί, να παρασχεθούν κίνητρα για την αποφυγή εκπομπών και για να γίνει αξιόπιστο για τους ενδιαφερόμενους τομείς. Πιστεύω πως έχουμε πολλά κλειδιά για να το κάνουμε πιο αποδοτικό. Αρχίζουμε με την φιλοδοξία, έχουμε υποσχεθεί μια μείωση διοξιδίου του άνθρακα κατά 40% τουλάχιστον. Οπότε το ETS πρέπει επίσης να βοηθήσει για να επιτύχουμε την τιμή αυτή των 40%. Και στον γραμμικό συντελεστή μείωση θα πρέπει να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά. Επίσης βλέπω πως πέραν από το ETS και άλλοι τομείς πρέπει να συνεισφέρουν θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Το ETS και το μη ETS. Αναγνωρίσαμε πως οι συγκοινωνίες είναι ένας τομέας με αυξανόμενες εκπομπές. Αναφερόμασταν έως στιγμής στις εναέριες μεταφορές, επίσης θέλουμε να συμπεριλάβουμε την αυσιπλοεία και υπάρχει και συζήτηση γιατί να μην συμπεριλάβουμε και τις οδικές συγκοινωνίες θα ήταν πολύ εύκολο να αναφερθούμε επίσης στα καύσιμα και να φροντίσουμε για εισφορές από τα καύσιμα. Αλλά αποφασίσαμε αλλιώς πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τις οδικές συγκοινωνίες. Αλλά αυτό είναι μια έλλειψη. Πώς ασχολούμαστε μόνο με τη βιομηχανία και όχι τη συγκοινωνία και τα κτίρια με, τις τις... με τα καύσιμα για θέρμανση. Αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε. Τώρα. Στο μέλλον ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε πως το ETS μπορεί να συμπεριλάβει και άλλους τομείς. Τώρα, εντός του ETS είμαι επίσης υπέρ μιας ακριβέστερης κατανομής των δωρεάν δικαιωμάτων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης, όπου μπορεί να μπει ο καθένας και να πάρει τα δωρεάν δικαιώματά του. Πιστεύω πως πρέπει να περιοριστεί το φαινόμενο στους τομείς οι οποίοι το χρειάζονται λόγω της κατάστασής τους στον ανταγωνισμό. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε πόσες βαθμίδες θα εισάγουμε. Η προσέγγιση με περισσότερες βαθμίδες είναι ίσως επίσης μια δυνατότητα. να αντιμετωπιστεί η διαφορετική ανταγωνιστική ένταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Και ως προς τους δείκτες αναφοράς πιστεύω πως επίσης μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια καλύτερη βαθμίδωση, διαβάθμιση. Ίσως από το 0,3 μπορούμε να πάμε στο πάνω από το 1,5. Επειδή διαφορετικές εγκαταστάσεις και διαφορετικοί τομείς έχουν επίσης διαφορετικές ανάγκες κατά την επόμενη δεκαετία. Άκουσα πολλές εκδηλώσεις Χρειαζόμαστε ρίζοσπαστική τεχνολογία σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάρη στη χημεία, στα λιπάσματα, στο τσιμέντο, στο χάλιβα, στα μη σιδηρούχα μέταλλα. Και το ερώτημα είναι ποιος θα καταφέρει το άλμα από τις σημερινές βιομηχανικές διεργασίες σε αυτές χωρίς ή με λίγες εκπομπές. Και αυτό το άλμα στην επόμενη δεκαετία θα κοστίσει πολλά χρήματα. Εδώ είναι που ελπίζω πως θα ενισχυθεί το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο δεν αρκεί για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να συνεισφέρουν και άλλοι, όπως το Ταμείο Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό του. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα πακέτο. για να μετατρέψουμε τα πρωτότυπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εμπορικά χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα επαναστατικό άλμα σε κάποιους κλάδους. Και εκεί πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα κονδύλια από το ETS. Ναι, κάποιες περιφερειές πληγούν ισχυρότερα από άλλες. Πρέπει να σκεφτούμε την κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Πιστεύω πως ένα ταμείο κοινωνικής δίκαιης μετάβασης, το οποίο θα μπορέσει να πάρει κονδύλια από το ΤΙΕΣ, θα ήταν ένα μήνυμα προς δήμους ή περιφέρειες, αλλά και στους κατοίκους, πως δεν τους αφήνουμε μόνους τους, αλλά βοηθούμε. Έχουμε κάποιες τροπολογίες, τις οποίες θα καταθέσουμε και ελπίζουμε πως στην ψηφοφορία των σκιωδών θα επιτύχουμε μεγαλύτερες πλειοψηφίες. Ο φάκελος αυτός δεν μπορεί να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο με οριακές ψηφοφορίες, επειδή ξέρουμε πως το Συμβούλιο θα πριονίσει και πάλι όλες τις φιλοδοξίες μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ευρείες, πληρο, ευρείες πλειοψηφίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Γκρουσίπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ολόθερμα τον Ιαν ε, Ντάνκαν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλε. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και διαπιστώνουμε και ε, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν για ε, τις χώρες οι οποίες ε, θα τιμωρηθούν με το νέο σύστημα, για να τα πω έτσι, σε οικονομικό επίπεδο λόγω του συστήματος αυτού. Η διαδικασία τώρα να ακολουθήσουμε διαφορετικές τεχνολογίες επιστήρει ένα μεγαλύτερο κόστος. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για αυτές τις διαδικασίες εξυγχρονισμού. Θα ήθελα όμως να τονίσω πως ε, σε κάποιους τομείς, όπως ε, ο τομέας παραγωγής γύψου, παραδείγματος χάρη, έχει εξυγχρονιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διαθέτουμε πλέον ε, προηγμένες τεχνολογίες, όμως δεν οφείλεται μόνο δεν οφείλονται οι εκπομπές μόνο στα καύσιμα, αλλά σε κάποιες ε, χημικές διεργασίες που ε, διαπιστώνουμε ότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές. Είναι όμως ε, αναστρέψιμες εκφύσεως αυτές οι διεργασίες και ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτή την πτυχή και να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας σε αυτό το τομέα για να αποφύγουμε τη διαρροή άνθρακα. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ένα άλλο σημείο. Η βιομηχανία θέρμανσης σε χώρες με μακρύ χειμώνα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι υπάρχουν ε, πηγές θέρμανσης με χαμηλές εκπομπές σε πολλές πόλεις ε, ε, στη χώρα μου, μεταξύ άλλων. Η βιομηχανία θέρμανσης λοιπόν ε, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές, ε, υπό την προϋπόθεση φυσικά θα λάβει και την απαιτούμενη στήριξη ο κλάδος αυτός. Βλέπουμε λοιπόν θετικές τάσεις ε, για τις ε, δημοτικές υποδομές ε, θέρμανσης, παραδείγματο που καλύπτονται από το ETS, ε, ενώ πηγές θέρμανσης χαμηλών εκπομπών έχουν αποκλειστεί από το σύστημα. Θα έπρεπε λοιπόν ενδεχομένως να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να κατευθυνθούν προς αυτές τις δημοτικές μονάδες θέρμανσης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Είναι πολύ μεγάλο το δυναμικό ε, της ε, ε, συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος βάσει των υπολογισμών που έχουν γίνει στην Πολωνία. Ο κλάδος θέρμανσης, εάν λάβει την κατάλληλη στήριξη, θα μπορούσε να προσφέρει 6 με 7.000 ΜΒ Εάν όμως λάβει χρηματοδότηση, ξαναλέω, από το Ταμείο ε, σου ούτως ώστε να περάσουμε από την ε, αποκλειστική παραγωγή θερμότητας στη μεικτή, στη συμπαραγωγή ε, θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος. Νομίζω ότι σε αυτή την νέα πρόταση θα έπρεπε να ε, λάβουμε υπόψη και τέτοιου παράγοντε όταν εξετάζουμε την μελλοντική νέα αρχιτεκτονική του ETS. Πολλοί συνάδελφοι επέστησαν την προσοχή μα στο Ταμείο Καινοτομία και στη χρήση αυτού. Αφενός μιλάμε για την ε, έστω και μερικά λήψη των ε, τομέων που έχουν προς το παρόν αποκλειστεί από το σύστημα ΙΤΕΣ για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ξαναλέω, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος οδηγεί σε πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, το επιδιωκόμενο δηλαδή. Τρίτον, ε, τον έφερε ο Τσέχος συνάδελφος. οι βιοτεχνολογίες και η δέσμευση άνθρακα. CCS ε, είναι πολύ ακρίβες αυτές οι νέες τεχνολογίες, όμως ε, κρύβουν ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Με καλή εφαρμογή της νομοθεσίας ε, και αξιοποίηση του δυναμικού δέσμευσης άνθρακα, μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ο τομέα εξελίσσεται διαρκώς και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχετικές συστάσεις Συμφωνία του Παρισιού. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα αυτά που ε, στοχεύουν συγκεκριμένα τα εργοστάσια. Για την ε, μόλυνση των εδαφών είναι δύσκολο ζήτημα, το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να στοχεύσουμε ε, τις καλλιεργητικές μεθόδους ε, που αποσκοπούν στην ε, παραμονή των φυσικών λιπασμάτων μέσα στο έδαφος. Θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τέτοιες καλλιέργειες κατά τη διαστολή με άλλες που οδηγούν σε πολύ μεγάλη διαρροή οργανικών ουσιών από το έδαφος. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για να ληφθεί αυτό το δεδομένο υπόψη, όμως διαπιστώσαμε ότι ε, σε περιπτώσεις όπου το έδαφος είχε χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς ε, σκοπούς και είχε διαβρωθεί, μπορέσαμε να ανακτήσουμε ένα μέρος αποτελεσματικότητας ε, του εδάφους. Σας ευχαριστούμε, κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω βεβαίως αυτό που ανέφερε ο συντονιστής ε, της ομάδας, την, πολιτική ομάδα στην οποία συμμετέχω, αλλά θέλω να επανέλθω σε δύο σημεία. Καταρχήν λυπάμαι που υπάρχει αυτή η προσέγγιση η σταδιακή, διότι αυτή οδηγεί σημαντική μείωση των δωρεάν ποσοστώσεων για κάποιου τομεί που περνάνε από 100% σε 50% ποσόστοση ε, και αυτό σε μια στιγμή όπου η κατάσταση για τη μείωση των εκπομπών αλλά και στο πλαίσιο του διεθνού, ανταγωνισμού, ανταγωνισμού, δεν έχει αλλάξει τόσο δραματικά. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένας πραγματικός κίνδυνος απώλειας ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας σε σχέση με την, τον υπόλοιπο κόσμο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται σαφώς βέβαια, αλλά αποτελεί αντικείμενο ε, συζήτησης δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τι γίνεται με, ε, με το benchmark για, για την ε, ζέστη, για την ε, θερμότητα. Ε, για να πετύχουμε τους στόχους του OTS, η παραγωγή εκπομπών που προέρχονται από τη βιομάζα δεν υπολογίζονται. Δεν νομίζουμε αυτό το σύστημα να συνάδει με το, παράγον, με το, με υπάρχον σύστημα παραγωγής. Μπορεί να είναι μια λύση αυτή για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για μεγάλους τομείς εντατικής παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κριτήρια ε, βιωσιμότητας που να ε, προσαρμόζονται στις υπάρχουσες σπόρους, στις ιδιαιτερότητες. Δεν πρέπει αυτό να είναι πιο επιζήμιο από το ίδιο το φυσικό αέριο. Το να μεταφέρει κάποιος δηλαδή βιομάζα επί πολλά χιλιόμετρα και αυτό είναι παραγωγή εκπομπών. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε, συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν συμμετείχα στην παρουσίαση, δεν ήμουν εδώ στην παρουσίαση της έκθεσης από τον κύριο Ντάνκαν, αλλά ήθελα να σας παρουσιάσω τις πρώτες μας αντιδράσεις. Εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός την πρωτοβουλία του να οργανώσει τεχνικές ε, ε, ακροάσεις γιατί είναι εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα και αυτές οι ακροάσεις είναι χρήσιμες. Επίσης εκτίμησα ιδιαίτερα την πρώτη του πρόταση αύξηση δηλαδή της ε, γραμμικής ε, παραγωγής, της γραμμικής μείωσης, συγγνώμη, ε, ξέρουμε ότι το 2,2% του LRF ε, αρκεί ίσα ίσα για να πετύχουμε τους στόχους της μείωσης του 40% στο 2030. Έτσι λοιπόν αυτό δεν αρκεί για να εγγυηθούμε τη μείωση τη τάξης των 90% στο 2050. και για να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας. Θα χρειαστεί λοιπόν μια πιο ε, έτσι, θαραλέα στάση και θα προτείνουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν συμφωνούμε με την ιδέα της αύξησης του κατοφλίου για τους μικρούς ε, εκπομπής, αν θέλετε. Ε, και η ανάλυση του κινδύνου ε, σε ό,τι αφορά την απώλεια άνθρακα, την διαρροή άνθρακα, από αυτά που έχουμε δει πρόσφατα, ακόμα και με μια τιμή 40-55 ευρώ το ανατόνο, είναι αρκετά ε, δύσκολο να υπάρξουν σημαντικές αποκλήσεις, σημαντικές διακυμάνσεις. Οπότε δεν συμφωνούμε με αυτό το μέτρο. Συμφωνούμε όμως να επανεξεταστεί το κατόφλι. σε ό,τι αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων για να αποφύγουμε αυτά τα windfall profits. Συμφωνούμε επίσης να υποστηρίξουμε το Ταμείο για την Καινοτομία μόνο χάρη στην καινοτομία και χάρη στην πραγματική μείωση των εκπομπών μπορούμε να ελπίζουμε να μειωθεί η πίεση. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αυτό με έναν απλό μηχανισμό πληρωμών ε, για τις άδειες εκπομπών. Έτσι λοιπόν ε, η καινοτομία για να βρεθούν καλύτερες τεχνολογίες ε, σε ό,τι φορτιστά να με ενέργειας είναι πολύ σημαντικές και δεν είμαστε καθόλου υπέρ του CCS. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η κατανομή των κονδυλίων να συνδέεται άμεσα με το πόσες εκπομπές μπορέσαμε να μειώσουμε. έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η οδηγία να πετύχει τον στόχο της. Την μείωση δηλαδή ε, της εκπομπής αερίων που προκαλούν το θερμό του θερμοκηπίου. Ε, θα υποβάλουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίες έτσι ώστε αυτή η οδηγία να σεβαστεί τον βασικό της στόχο. Ιδάλλως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, δεν θα είναι αποτελεσματική και θα οδηγήσει και σε απάτη και σε κερδοσκοπία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε αυτό το εργαλείο να λειτουργήσει καλά, ορθά Ιδάλλως κινδυνεύουμε να μην πετύχουμε τους στόχους μείωσης που έχουμε θέσει. Θα το δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θα ήθελα να θυμίσω πως σήμερα έχουμε χάσει πολλούς συναδέλφους διότι συνεδρία ταυτόχρονη η Επιτροπή εμείς ε, για τα, τις εκπομπές των αυτοκινήτων. και ε, έχουν πάει σε εκείνη τη συνεδρίαση γιατί είναι υπεύθυνοι πολλοί συνάδελφοι για φακέλου σε εκείνη την επιτροπή. Εμείς, εμεί είπα. Ειδική Επιτροπή για τι εκπομπέ των αυτοκινήτων. Ο κύριος ε, Ντάνι Μίτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντάνκαν, για την έκθεσή του ε, και για τι εντατικέ διαβουλεύσει που έκανε με του συναδέλφου του τελευταίου μήνε. Ε, νομίζω ότι φαίνεται αυτό που προκύπτει από τη σημερινή συζήτηση. Καλωσορίζουμε την έκθεση και από ό,τι βλέπουμε από τα σχόλια των βουλευτών, η πρότασή μας πρόταση που κατατέθηκε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ε, πέρυσι ε, έχει ως στόχο ε, να δώσει συνέχεια συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2014 αρχικά και εάν οι συνομοθέτες επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να το επιτύχουμε. Ε, όμως η πρότασή μας συνάδει με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014 ε, αναφέρθηκαν πολύ στη Συμφωνία του Παρισιού και τη σημασία της. Ε, το ETS δεν είναι το μόνο μέτρο, το μόνο μέσο που προτείνουμε. Την, περασμένη, την προπερασμένη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, πρότεινε Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση επικύρωση Συμφωνία του Παρισιού και θέλουμε ε, να προωθηθεί αυτή η συμφωνία από αυτή τη πρόταση. Ε, μίλησαν πολύ για την πρόταση για το effort sharing και για τη χρήση γης ε, για τη γεωργία και θα καταθέσουμε σχετικές νέες προτάσεις πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σχολιάσω τρία-τέσσερα από τα σημεία που ήγηραν οι συνάδελφοι και να προσπαθήσω να απαντήσω ε, αμέσως μετά στις ερωτήσεις που μας απευθύνατε. Great. Firstly... Πρώτα απ' όλα, για το Παρίσι για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι κέρια σημασία η αίσια λειτουργία του ETS. Η Κίνα, η Κορέα εκπονούν ε, αντίστοιχα συστήματα για την τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θα πρέπει εγκαίρως να φροντίσουμε να λειτουργήσει το ETS. Για τα benchmarks, επειδή τονίστηκε η σημασία τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει μια πρόταση βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα για την ε, ουσιαστική κατανομή των ποσόστων ε, στο 10% των πλέον επιτυχημένων αποτελεσματικών υποδομών βάσει και της πρώτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας. Η διαδικασία συναπόφασης και όχι σε διαδικασία επιτροπολογίας αποφασίζονται αυτά. Νομίζω ότι είναι βασικό αυτό το στοιχείο. Ε, ο εισηγητής ε, προτείνει να έχουμε επιπρόσθετους ε, συντελεστές Επιπρόσθετου ποσοστό. Ξαναλέω, βασιζόμαστε σε πραγματικά δεδομένα για να δούμε ακριβώ η κλάδοι ποια αύξηση αποτελεσματικότητα έχουν επιτύχει για τις ε, προηγμένες τεχνολογίες breakthrough και την ε, χρηματοδότηση για την ε, καινοτομία. Φυσικά είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν στην αγορά αυτές τις τεχνολογίες, να βγουν από το τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να χρησιμοποιηθούν στην αγορά. Και εκεί θέλουμε, χρειαζόμαστε από, πραγματικά αυτά αποτελέσματα και χαίρομαι που το τονίσατε κι εσείς. Επίσης, ανανέωση της δυνατότητας opt-out για τους small τους, ε, τις μικρές εγκαταστάσεις. Ε, το αναφέρουμε στη νέα μας πρόταση και ε, γιατί, διότι θέλουμε να έχουμε την, μια ισορροπία, να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Και τέλος, η χρήση των εισοδημάτων από το σύστημα. Τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής έχουν πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποιούν το 90% των εισοδημάτων από το ETS για την, τα μέτρα μέτρα αντιμετώπισης και προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Ε, υπάρχει μια υποχρέωση σε soft law ε, για να χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα για αυτό το στόχο. Πέρυσι τον Ιούλιο ένα μέρος πρότασης μας ε, περιστρεφόταν γύρω από αυτό, χρήση του εισοδημάτων για την χρηματοδότηση της μετάβασης. Φυσικά έχουμε επίγνωστο ότι χρειάζεται αυτή η μετάβαση και γι' αυτό έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό. Περνώ στις ερωτήσεις. Ο κύριος Πόξ μας είπε πώ καταλήξαμε στο 57% με ποιο υπολογισμό. Νομίζω δεν θα ευσέλθω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να σας πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε γραπτές απαντήσεις ακριβώς ε, για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του 57%. Ξέρω ότι έχουν κυκλοφορήσει και άλλοι τρόποι υπολογισμού. Θα ρωτήσω τους συναδέλφους μου και θα δω αν μπορώ να σα στείλω αυτόν τον ε, τρόπο υπολογισμού που στείλαμε στα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε και στην ε, δασοκομεία. Ε, φυσικά συμφωνούμε εμείς στην Επιτροπή ότι όλοι οι κλάδοι πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και αυτό είναι και μέσα στην πρότασή μα για την επικύρωση Συμφωνία του Παρισιού. Είναι διατομεακή η προσπάθεια. Για την δασοκομεία σα είπα πριν τις καλοκαιρινέ διακοπές θα καταθέσουμε πρόταση για την δασοκομεία για τη χρήση των εδαφών και τη συμβολή των τομέων στη μείωση των εκπομπών. Ε, το ίδιο και για τη βιομάζα, γιατί αναφέρθηκε και αυτό από τους συναδέλφους. Ε, για την θέρμανση και την αποτελεσματικότερη δημοτική θέρμανση, κυρίως σε αστικές περιοχές. Ε, στην πρότασή μας ε, αντιμετωπίζουμε όλες τις διαστάσεις ε, του προβλήματος και γι' αυτό ε, σωστά τονίσατε και στο το ρόλο των μηχανισμών χρηματοδότησης για να προωθηθεί η, δημόσια θέρμανση, η δημοτική θέρμανση τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν προτάσεις για την μείωση των εκπομπών εκτός ETS, όπως αυτές προέρχονται, ε, εκπομπές προέρχονται από την θέρμανση των σπιτιών. Νομίζω ότι κατά ε, την ε, αναθεώρηση των μέτρων που έχουν προκύψει από το Παρίσι θα συνεχιστεί η συζήτηση και αυτό θα συμπεριληφθεί στα μέτρα που θα σας υποβάλουμε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Λάβια, ευχαριστούμε. Ε, ήθιστε να ακούμε τον εισηγητή μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει τη συζήτηση, όμως ε, ο συνάδελφος μας ε, μας ζήτησε ειδικά να κάνουμε μια εξαίρεση, διότι ήταν σε αυτή την επιτροπή μας. Εγώ θα του δώσουμε το λόγο και μετά στον κύριο Τάνικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που άργησα. Η καθυστέρησή μου οφείλεται σε υποχρεώσεις που είχα στο Κοινοβούλιο Πιστεύω πως θα μπορέσω να προσπαθήσω να αντιδράσω σε αυτό που υπόθηκε αν και δεν το άκουσα προσωπικά. Αλλά πιστεύω πως μπορώ να διασανθώ τι κάνει ο κύριος Ντάνκαν. Για την πρώτη παρατήρηση, τη στρατηγική του κυρίου Ντάνκαν. Λέει πως δεν είναι τόσο αυτό που περιμένω αυτό που θα, σε αυτό που θα καταλήξουμε. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στρατηγική, επειδή όλοι γνωρίζουμε πως η, βάση of industry to try to dilute. Για μια έκθεση Denvi είναι πάντα το σημείο από το οποίο προερχόμαστε. Και τότε από την Επιτροπή αυτή πηγαίνουμε στην Ολομέλεια, έχουμε τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Πότε δεν υπόθηκε πως η Envy θα συζητήσει με το Συμβούλιο. Δηλαδή η στρατηγική του κυρίου Τάνκαν, αν είναι αυτή, τότε πιστεύω πως είναι ασφαλμένη επειδή θα έχει χαμηλότερα αποτελέσματα από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και πιστεύουμε πως ο κύριος Ντάγκαν κάνει ένα στρατηγικό σφάλμα τώρα. Θα εξηγήσω σύντομα γιατί μιλούμε για μια έκθεση χωρίς την παραμικρή φιλοδοξία. Ο κύριος Ντάγκαν είναι πάντα πολύ περήφανος για την τριπλή φιλοδοξία του. Πρώτα απ' όλα λέει πως επιφανειακά πρέπει να κοιτάξουμε αλληλοεπικαλυπτόμενες πολιτικές. Αυτό που εννοεί όμως είναι ότι επιτυχείς πολιτικές όπως η οδηγία περί ανανεώσιμων δεν θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί επειδή τα καταραμένα τα ανανεώσιμα μειώνουν τις εκπομπές σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή ότι πρέπει να παρατηθούμε από μια λειτουργική πολιτική για να λειτουργήσει το ETS. Και θα έλεγα πως αυτό είναι ο λάθος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Επειδή αν θέλει κανείς ένα λειτουργικό ETS θα πρέπει να κοιτάξει τις αλληλοεπικαλυπτόμενες πολιτικές, αλλά να κάνει λειτουργικό το ETS. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Το δεύτερο, οι χώρες ε, ίσως αποσυρθούν από μια υπερπροσπορά δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι μια φιλοδοξία, αυτό είναι ένα ίσως. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που ίσως κάνουν οι χώρες, αλλά δεν το κάνουν. Αυτό δεν είναι φιλοδοξία, κύριε Ντάνκαν. Αυτό δεν είναι παρά μια ωραία διατύπωση. Και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τα οποία υπόθηκε ότι ίσως γίνει μια αναθεώρηση αργότερα, η οποία τοποθετήθηκε το 2023. Δηλαδή πιο μακριά στο μέλλον. Και όλοι γνωρίζουμε τι θα πει η βιομηχανία. Μην αλλάξετε τους κανόνες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και ο αγώνας είναι διαρκής. Οπότε ποτέ δεν μας επιτρέπεται να αλλάξουμε τους κανόνες. Το 2023 ίσως να μην βρίσκεστε εδώ. Ίσως και όχι μετά την Πέμπτη. Αλλά τότε έτσι αναβάλουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση σε άλλους οι οποίοι θα πρέπει να καταπολεμήσουν τα ίδια λόμπι όπως εμείς και πιστεύω πως εδώ έχουμε μια έλλειψη φιλοδοξιών και όντως έχω και κάποιες προτάσεις επειδή από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ ΕΛΚ και ECR πως όταν μιλούμε για τους δείκτες αναφοράς πρέπει να πάμε στις πραγματικές εκπομπές. Εντάξει, αν οι πραγματικές εκπομπές είναι τόσο σημαντικές, ας αρχίσουμε τότε με το 2021 με βάση τις πραγματικές εκπομπές. Επειδή γνωρίζουμε πως η Ευρώπη πληρεί τώρα το 27% των εκπομπών. Δηλαδή αν παίρνετε τόσο στα σοβαρά τις πραγματικές Εκπομπε, τότε α έχουμε και μια ημερομηνία αναφορά, Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι μιλούμε μόνο για δείκτε αναφορέ, αλλά και όχι για ημερομηνία αναφορά. Αναμένω λοιπόν μια κάποια συνέπεια από εσά, κύριε Ντάνκαν. Δηλαδή τη ημερομηνία αναφορά για την αλλαγή τη του ETS. Ε ε, ε, μετά, οι συντελεστέ γραμμική μείωση. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτε, υπάρχουν περιθώρια αύξηση των γραμμικών συντελεστών. Ακόμα και στο Συμβούλιο χτε κάποιε χώρε είπαν πω πρέπει να αυξηθούν. Ο κύριο Ντάνκαν λοιπόν θα είναι βοηθό στη συζήτηση εκείνη ή θα την καταπνίξει πριν καν αρχίσει. Και πιστεύω πω ω Επιτροπή ΕΝΒΗ πρέπει να τοποθετηθούμε υπέρ τη συζήτηση. Και η πρόταση 2-2 δεν θα φέρει όλη την, την ευρωπαϊκή οικονομία στα μείον 80% το 2050. Ούτε καν το σενάριο των 2 βαθμών Κελσίου θα επιτευχθεί. Αυτό δεν συμμορφώνεται με το, τους στόχους του Παρισίου και δεν χρειάζομαι μια συνεδρίαση το 2023. Οπότε, μια μετριοπαθής πρόταση, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε οι, οι γραμμικοί συντελεστές να είναι εναρμονισμένοι με το, με το σενάριο ως προς τη θερμοκρασία η πιθανότητα να ξεπεράσουμε τους δύο βαθμού θα έρχεται στο 1 τρίτο. Αυτό συζητούμε εδώ. Αυτό είναι πολύ μετριοπαθέ από του πράσινου και είμαι σίγουρο πω και άλλοι θα πούνε ότι παρά είμαστε μετριοπαθεί εδώ. Όσον αφορά το Ταμείο Καινοτομία. Είναι βασική σημασία. Ναι, η καινοτομία είναι σημαντική. Αλλά τι κάνει ο κύριο Ντάνκαν. Πρώτα απ' όλα μεταθέτει 150 εκατομμύρια μη δεσμευμένων πόρων στο ταμείο αυτό. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με αυτό. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν ήδη χρησιμοποίησε τα, τους μη δεσμευμένου πόρους που πάνε στο ΕΝΙΑΡ. E Και τώρα, εκτός από αυτό, εκτός από τα 150 εκατομμύρια που πάνε στο ΕΝΙΑΡ, e μείωση των θέλει να βάλει στην, στην καινοτομία, δηλαδή διπλά βιβλία. Γιατί χρησιμοποιούμε τα αχρησιμοποιητά δικαιώματα από την προηγούμενη φάση για την επόμενη. Γιατί το κάνουμε αυτό. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε το Ταμείο Καινοτομίας αυτό είναι εντάξει. Αλλά τότε γιατί να χρησιμοποιούμε αχρησιμοποιητά δικαιώματα από την προηγούμενη φάση. Είναι αχρησιμοποιητά, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάστηκαν, δεν ήταν αναγκαία. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε με σοφό τρόπο. Και το τελευταίο ζήτημα στη διάσημη συζήτηση για το κατά πόσον έχουμε αρκετά δικαιώματα δημοπράτησης ας είμαι σαφής αν υπάρχει ανάγκη για ένα διατομεακό συντελεστή διόρθωση τον οποίο όλοι θέλουμε να αποφύγουμε αυτό σημαίνει πως σπαταλούμε δωρεάν δικαιώματα σε τομείς που δεν τους χρειάζονται και επίσης στην πρότασή σας κύριε Τάνκαν δίνουμε 30% δωρεάν δικαιώματα σε τομείς που δεν έχουν διεθνή ανταγωνισμό. Εγώ νομίζω ότι τα διεθνή δικαιώματα δίνονται μόνο σε τομείς που έχουν προβλήματα με το διεθνή ανταγωνισμό. Γιατί λοιπόν δίνουμε δωρεάν τέτοια δικαιώματα, ας μην το κάνουμε λοιπόν. Και όσο περισσότερο διανέμουμε χωρίς τον παραμικρό λόγο δωρεάν, τόσο περισσότερο θα προκύψει η ανάγκη για έναν διατομιακό συντελεστή διόρθωσης. Και μην πούμε, αν αυτό χρειαστεί, θα χρειαστούμε περισσότερα δωρεάν δικαιώματα. Όχι. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα ελεύθερα δικαιώματα, τα δωρεά δικαιώματα να πηγαίνουν στους τομείς που τους χρειάζονται. Κάθε τομέα, αλλιώ θα πει θέλουμε περισσότερα ελεύθερα δικαιώματα. Όλοι μας θέλουμε. Αλλά κανείς δεν λέει ποιος τομέας δεν χρειάζεται ελεύθερα δωρεά δικαιώματα. Επειδή δεν το κάνουμε αυτό ως βιομηχανία. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο όλοι ζητούν όλο περισσότερα δωρεάν δικαιώματα. Στο τέλος θα έχουμε ένα λόμπι στο οποίο θα υπακούν οι πολιτικοί και θα δίνουμε όλο και περισσότερα δωρεάν δικαιώματα και στο τέλος θα καταλήξουμε σε έναν διατομεακό συντελεστή διόρθωσης. Γι' αυτό αν δεν το θέλετε αυτό, ας είστε λίγο πιο αυστηροί και ας τα χορηγήσετε μόνο στους τομείς που όντως τα χρειάζονται, αντί να τα δίνετε τζάμπα για όλους. Και αυτό σημαίνει μια προσέγγιση όχι από αυτή, σαν και αυτή που προτάθηκε από κάποιους συζητητές αυτή τη αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή κύριο Ντάγκαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευτυχώς που ήρθε ο Μπάς γιατί υπήρχε αρμονία. Είναι δύσκολο πάντως να επικρίνει κάποιος ε, ε, σχόλια τα οποία δεν άκουσε καν, έτσι. Συγγνώμη που θα επαναλάβω κάπως τον εαυτό μου, αλλά το πρώτο θέμα είναι ότι η οδηγία για το ανανεώσιμα έχει στεφθεί από επιτυχία, καθώς και η οδηγία για την αποδοτική χρήση ενέργειας. Δεν έχω εγώ την, πρόθεση να την ερώσω σε καμία περίπτωση. Αυτό που θα ήθελα όμως είναι να φύγουν οι δωρεάν ε, ε, ε, allowances στον τομέα της προσφοράς. Αυτό είναι το πρώτο. Εάν το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να δούμε όμως πόσο επιτυχής είναι αυτές οι πολιτικές και να τις σχετίσουμε μεταξύ τους. Είπε και ο κύριος Μπέρντ, δεν τα να ακούσετε ούτε αυτόν, ότι το θέμα να υπάρχει διάδραση και όχι επικάλυψη. Πώς θα οδηγηθ, μας οδηγήσουν αυτές οι πολιτικές και που θέλουμε να πάμε. Σε ό,τι αφορά την εθελοντική απόσταση είπα May, εντάξει, να το κάνω must το May, δεν έχω καμία επιμονή για το ΜΕΙ. Ένα κράτος μέλος έχει ως στόχο να θέσει τόσο υψηλούς στόχους, τότε πρέπει ε, να, το, να το τηρήσει το στόχο. Δεν μπορούμε πλέον να κοροϊδεύουμε. Πρέπει τα κράτη-μέλη αυτό που λένε να το εννοούν. Και αυτό σημαίνει ότι αν απελευθέσουμε ένα μεγάλο αριθμό allowances και ε, σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε εφόσον υπάρχει σημαντική κυριαρχία στα κράτη-μέλη. Ε, και τότε θα δούμε ποια, ποιο κράτος μέλος είναι φιλόδοξο και ποιος υπέγραψε μόνο έτσι επειδή τα είχε πιει λίγο, παραπάνω στο Παρίσι. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναθόρηση του 2023, αν περιμένω στο 2023, όντως θα έχουμε περιμένει πάρα πολύ. Α ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα. Το είπα και νωρίτερα. Όταν θα φτάσουμε το 2023 λοιπόν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι, όχι να τελειώνουμε, να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, η φιλοδοξία μου εδώ είναι να εξετάσουμε τον όγκο και όχι τη γραμμική μείωση και όχι το, ε, ε τον παράγοντα γραμμικής ε, μείωσης. Εάν μειώσουμε τον όγκο, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να προχωράμε. Ε, επίσης κάτι άλλο, ε, η ομάδα μου ετοίμασε μια πολύ σημαντική ομιλία για μένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο να πω κάτι που δεν είπα προηγουμένως, ότι μπορεί να βοηθήσει. Ε, εγώ δεν είμαι υπέρ του παράγοντα αυτή τη γραμμική μείωση. Πρέπει να εξεταστεί αυτό με βάση τι δεσμεύσει. Και είμαι έτοιμο να δεχτώ και να προτείνω ακόμα 2,4% ε, για τον παράγοντα αυτό, αν, αν αυτό μα οδηγήσει να προχωρήσουμε. Πρέπει να πετύχουμε του στόχου μα όμω ε, νομίζω χωρίς να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση το θέμα των unused allowances των δικαιωμάτων που δεν χρησιμοποιούνται. Ε, είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Λογικό μου φαίνεται. Ακούστηκαν και κάποια άλλα εξαιρετικά χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις. Ξέχασα και τους προηγούμενους και σίγουρα αυτά θα τα ενσωματώσω και θα τα συμπεριλάβω. Μπορούμε να φτάσουμε σε συνένεση, μπορούμε να πετύχουμε αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο σε ό,τι αφορά τώρα την ε, κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή εξετάζοντας το θέμα του όγκου μετά τη Συμφωνία του Παρισιού. Ε, εάν πρέπει να έχουμε υψηλότερο παράγοντα γραμμική μείωση θα το κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο. Εγώ δεν είμαι εδώ ως αυτός που λέει ότι υπάρχει βεβαιότητα για το τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ θέλω να συγκεράσω τις απόψει για να πετύχουμε το στόχο μας. Έχω δεχθεί επικρίσεις ε, και στα κοινωνικά μίντια επ' αυτού, αλλά εγώ επιμένω. Είμαστε δημοκράτε. Ε, εάν δεν σας αρέσει η έκθεσή μου, τροποποιήστε την. Αν θέλετε να αλλάξετε, αλλάξτε την. Ε, και αν βρείτε του ψήφου που χρειάζεστε θα αλλάξει. Έχουμε μια μικρή ομάδα. Εγώ ξανά και ξανά το έχω πει αυτό και κάτι ακόμα επειδή ε, είναι σημαντικό το θέμα των κοινωνικών μέσων. Προτιμώ έναν διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο από ότι να μου στέλνει κάποιο κόμικ ή κινούμενα σχέδια για να μου εξηγήσει τόσο περίπλοκο ζήτημα ε, ε, με, τον, με έναν Batman που δίνει ένα χαστούκι στο Ρόμπιν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και τα κόμικ και τα κινούμενα Δεν είναι κόμικ αυτή η υπόθεση. Είναι τεράστιε επιπτώσει αυτή τη υπόθεση. Δεν μπορούμε να τα σκεφτόμαστε κατακρεματισμένα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα νοσοκομεία, η νοσοκομεία πρέπει να αποτελέσει μέρο αυτού. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα. σω και να μην πρέπει να είναι ή να πρέπει να είναι. Κάποιο λέει γιατί να μην κάνουμε το ETS από τη μια πλευρά και το, το μη ETS από το υπόλοιπο, αλλά δεν είμαι εγώ αυτό που αποφασίζει την Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο μαζί. Απευθύνομαι σε όλου εδώ, όχι σε αυτού που είναι μόνο μπροστά μου και δεξιά μου και αριστερά μου και αυτού που είναι πίσω μου και η βοηθή, ε, η πολύτιμη συνεισφορά του δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Λοιπόν, ε, για να σημειώσουμε πρόοδο πρέπει να φανούμε έξυπνα, να φερθούμε έξυπνα όμω. Και θα επαναξετάσουμε το Παρίσι και θα πετύχουμε αυτό το 1-5 και αν το μπορέσω να το κάνω αυτό θα το κάνω. Ε, θα πρέπει να γνωρίσουμε βεβαίω ότι ο κλάδο, η βιομηχανία είναι μέρο του οικονομικού κόσμου. Το να πλεί κάποιο το αντίθετο είναι ε, πραγματικά ε, να ε, εθελοτυφλεί. Βλέπω ότι σιγά σιγά χασμουριέται ο πρόεδρο, ίσω να το παράκανα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε, θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα και καλύτερα εφόσον σημειώσουμε, ε, εφόσον ενώσουμε τι δυνάμει μα και προχωρήσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι σκιώδη συγγητέ, σα ευχαριστώ για την συνεισφορά σας. Πιστεύω πραγματικά ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε τη συνάντηση, να σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμίες, ε, 28 Ιουνίου στι 12 μπορείτε να υποβάλλετε πλέον τροπολογίες, που είναι η προθεσμία και η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα γίνει ε, τον Δεκέμβρη. Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο ε, στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στη Δεν Μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα το πρωί. Θα τα ξαναπούμε ξανά το απόγευμα. Θα ξαναπούμε το απόγευμα στις 3. Στις 3 έτσι. Θα θυμίζω ότι στις 3 έχουμε εδώ την, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, για να υπογράψουμε την συμφωνία μας. Ευχαριστώ.